Thank you, colleagues. Good morning. Καλημέρα συνάδελφοι. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, υιοθέτησή τη. Αν έχετε αντίρρηση, να μου το πείτε, αλλιώ την υιοθετούμε. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Έχουν κυκλοφορήσει τα πρακτικά. Προτείνω να εγκριθούν τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 4η Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία. Άρα εγκρίνονται και τα πρακτικά. Επόμενο σημείο, Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Μία μόνο. Για τα νέα μέλη της Επιτροπής μας, αν υπάρχουν σημεία που θέλετε να συζητήσει η Επιτροπή, παρακαλώ είτε πείτε τα σε μένα, είτε πείτε τα στον συντονιστή σας, για να τα, μας τα πει στη συνεδρίαση με τους συντονιστές. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να θίξετε κάποια θέματα, να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε αν θέλετε διερευνήστε τις δυνατότητες που έχετε. Πάμε τώρα στο σημείο 5 το σημείο που συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, τα έκτακτα μέτρα για το Brexit που θα επιτρέψουν στα ε, βρετανικά σκάφη να αλλιεύουν στα ευρωπαϊκά ύδατα, εάν τα ευρωπαϊκά σκάφη επιτρέπεται να αλλιεύουν στα βρετανικά ύδατα. Ουσιαστικά δημιουργείται μια βάση στα πλαίσια και τη ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, για το πώ θα γίνει αυτό, αλλά βεβαίω σε περίπτωση που όντω γίνει το Brexit εξαρτάται από τι δύο ε, ε, πλευρέ και το κατά πόσο θα εξεύρουν μια συμβαστική λύση. Η πρόταση αυτή μπορεί να εγκριθεί από την απλουστευμένη διαδικασία χωρί τροπολογία σύμφωνα με τον, με τον κανόνα 52.1, ο οποίο έχει τύχει στήριξη από του συντονιστέ στην πρωινή συνεδρίαση. Η ομάδα εργασία Ελία του Συμβουλίου επίση ε, πρότεινε στην ΚΟΡΑΠΕΡ να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή χωρί ε, ουσιώδει αλλαγέ. Οπότε ρωτώ, τα μέλη αν μπορούμε να εγκρίνουμε τον ε, κανονισμό αυτό με την εμπιστευμένη διαδικασία χωρί τροπολογίε σύμφωνα με τον κανόνα 52. Πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσει. Κύριε Μοντή, θέλετε να μιλήσετε. Ναι. Δεν είμαστε αναπληρωματικά μέλη. Απλώς ήθελα να πω. Ε, ναι, να πω ότι επισήμω έχουμε αντίρρηση. Έχουμε καταστήσει σαφή τη θέση μα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολλή δρόμο ακόμα, ακόμα να διανύσουμε πριν να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε αμοιβαιότητα. Τώρα για να... αυτό το σημείο δεν μπορούμε να το στηρίξουμε σίγουρα. Ε, εντάξει. Ευχαριστώ. Ε, δεδομένου του ότι πρέπει να συμφωνήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν την καταλαβαίνω εδώ στη θέση σα, αλλά βεβαίω κάθε αντίρρηση είναι θεμητή. Άλλε αντιρρήσεις υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, 10% των μελών της Επιτροπής πρέπει να έχει αντίρρηση. 10% σημαίνει τρία μέλη. Άρα, μπορώ παρακαλώ να δω ποιες είναι, πόσες είναι οι αντιρρήσεις που έχουμε. Ο κύριος Μοντή έχει αντίρρηση, όπως είπαμε. Δύο. Άλλος υπάρχει. Είναι πάνω από δύο οι αντιρρήσεις. Δεν βλέπω πάνω από δύο. Επομένως πρέπει να υπάρχουν τρεις. Άρα για να... Αν η κυρία Ντότζ είναι εδώ, κάποιος από τους δυο σας που ήσασταν πραγματικά μέλη θα χάσει την ψήφο του. Λοιπόν, δύο αντιρρήσεις βλέπω όλες και όλες, άρα κάτω από 10%, άρα εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Κλείνουμε το σημείο αυτό. Το αν θα υπάρξει διαφορά θα εξαρτηθεί από το Brexit και τη συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση και βασιλιού μετά από αυτό. Πάμε στο σημείο 7. Το πρώτο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Το σημείο αυτό έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί προς το παρόν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία. Τα νέα μέλη μπορεί να μην το έχετε υπόψη σα το ταμείο αυτό, αλλά βεβαίω έχουμε και συναδέλφου που έπρεπε να το δημιουργήσουν, να το διαχειριστούν το ΕΤΘΑ, οπότε έχουν ε, ιδιαίτερη γνώση να μοιραστούν μαζί μας. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κυρία Ελίζα Βολάρη. Κομισιόν, έχετε το λόγο. Thank you, Good morning, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Έχω μια παρουσίαση PowerPoint, μπορείτε να τη δείτε. Θα καλύψω κυρίως ε, τα τρέχοντα για την ε, εφαρμογή και θα πω και λίγα ε, πράγματα για την πρόταση της Επιτροπής για το μέλλον. Το τρέχον ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έχει προκοδοτηθεί με 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 89% αυτών, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα, το διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη μέσω μεικτής διαχείριση. 11% το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμυγό για διάφορε δραστηριότητε, επιστημονικέ γνωμοδοτήσει, συλλογή δεδομένων, ε, η μπλε ανάπτυξη, θαλάσσια πολιτική, θαλάσσια ασφάλεια. Και βλέπετε εδώ και το, τα γραφικά για το πού πάνε τα διάφορα τμήματα του προπολογισμού. Το έτθα τώρα με δύο λόγια. Καταρχάς επικεντρωνόμαστε στους βασικούς στόχους της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Υιοθετήθηκε λίγο πριν τη μεταρρύθμιση το 2013, οπότε επικεντρώνεται όχι μόνο στην ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση και την μετάβαση στις βιώσιμες, στη βιώσιμη αλίευση, την υποχρέωση για τις εκφορτώσεις, αλλά και κάτι άλλο που είναι σημαντικό να πω, επικεντρώνεται και στην εξασφάλιση τη ε, οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, ένα καλό επίπεδο διαβίωση για του αλληλεί, κοινωνικά θέματα όπω α πούμε ασφάλεια επί του σκάφου, ε, συνθήκε εργασία για του αλληλεί, γυναίκε στην αλληλεία και γενικότερα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των αληφτικών κοινοτήτων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Βεβαίω, έχουμε μια ισχυρή πράσινη διάσταση σε ό,τι αφορά την προστασία τη βιοπικιλότητα, του Natura 2000. Έχουμε πολύ καλά project ε, όπου καταβάλλονται χρήματα στους ε, αλληλείς για να προστατεύουν τέτοιου είδους ε, περιοχές ή για να συλλέγουν θαλάσσια απόβλητα. Όπως είπα και πιο πριν, επικεντρωνόμαστε και στις τοπικές κοινότητες μέσω διαφόρων ε, τοπικών ε, εξελίξεων που τις διαχειρίζονται οι ίδιες οι κοινότητες. Συνεχίζεται δηλαδή αυτό που είχαμε ξεκινήσει το 2007 και το 2013 αυτές τις περιόδους. Έχουμε πάνω από 300 ε, ομάδες τοπικών αλλιέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε βεβαίω χιλιάδε project που τρέχουν. Όπω είπα πριν, έχουμε και μια ισχυρή ε, ε, στόχευση στην συλλογή δεδομένων και στον έλεγχο τη αλληλεία. Αλλά η κοινωνική στόχη τη κοινή ελευθερική πολιτική είναι επίση σημαντική. Δύο λόγια θα ήθελα να πω και για αυτού. Το Ταμείο ε, ευθυγραμμίζεται ως προς αυτούς τους στόχους και αυτό που βλέπουμε είναι τα κράτη-μέλη στα επιχειρησιακά τους προγράμματα να προσπαθούν με τη χρήση του Ταμείου, με τη βοήθειά του, να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου, που είναι η, ε, ο εμπλουτισμός των αποθεμάτων, ε, βλέπετε σε παρενθέσεις προσπαθούμε να στηρίξουμε τους νέους αλληλείς για να μπορούν να αγοράσουν ας πούμε το πρώτο του σκάφος, ένα σκάφος από δεύτερο χέρι μεταχειρισμένο για να τους επιτρέψουμε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, τους δίνουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσπαθούμε, έχουμε δυνατότητα να τους καταρτήσουμε, κάνουν ε, εταιρικέ σχέσεις με ε, επιστήμονες, οπότε υπάρχουν πολλά κονδύλια τα οποία διοχετεύονται στην αντιμετώπιση της ανανέωση των γενεών. Ε, ε, κάθε φορά βλέπουμε βεβαίω και ένα 1-2% απώλεια ε, κάθε χρόνο. Επίσης, μεγαλύτερε επενδύσεις στις ασφαλείς ε, συνθήκες εργασίας, ας πούμε, τουαλέτες, κουζίνες, ε, βαφές που δεν γλιστρούν, αντιολισθητικές. Οπότε όλα όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω στο σκάφο μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο. Και αυτό υπάρχει και στην πρόταση για το μελλοντικό Ταμείο. Η πτυχή του φίλου επίσης είναι πολύ σημαντική. 14% όλων των κοινοτήτων και των ε, σχετικών project που τα διαχειρίζονται οι κοινότητες ε, τα διαχειρίζονται οι γυναίκες και ο ρόλος των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη την αλυσίδα. Εδώ τώρα στην οθόνη βλέπετε το πώς διοχετεύονται τα κονδύλια. Βλέπουμε από αριστερά οι μπλε κολόνε, βλέπετε τι έχει προγραμματιστεί, οι μπλε στήλε, στα αριστερά βλέπετε τι έχουμε δαπανίσει για την αλληλεία, περίπου 1,6 δι ευρώ δηλαδή άμεσα για την αλληλεία, που περιλαμβάνουν και την κοινωνική διάσταση, όπω σα την ανέφερα πιο πριν, τις συνθήκες εργασίας επί του σκάφου, προσωρινέ παύσει, δηλαδή ε, πληρώνουμε του αλληλείς ε, που πρέπει να σταματήσουν για κάποιο λόγο να αλλιεύουν για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό επίπεδο διαβίωση, κατάρτιση κλπ. Μετά, δεύτερη στήλη, ότι δαπανούμε για την υδατοκαλλιέργεια. 1,2 δις ευρώ έχουν προγραμματιστεί να δαπανηθούν στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Και έχουμε τη συλλογή δεδομένων και, τον ελέ... τους ελέγχους. 1,1 δις ευρώ πάνε σε δραστηριότητε συλλογή δεδομένων και ελέγχου. Μετά έχουμε τα τοπικά ε, project από τι κοινότητε. Στα πλαίσια του UP5 έχουμε ε, στήριξη και για την ε, επεξεργασία, στηρίζοντα και τι δραστηριότητε θέσει εμπορία από του αλληλεί, για τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα κτλ. Το UP6 επίσης, ε, η προτεραιότητα δηλαδή είναι η αλληλευτική πολιτική και υπάρχει και η τεχνική βοήθεια, τεχνική αρρωγή που ενισχύει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους. Εδώ βλέπετε μία έτσι, γενική θεώρηση, δεν θα σας πω πολλά, αλλά βλέπετε εδώ ανά κράτος μέλος τι έχει προγραμματιστεί, πόσες, ε, ε, πόσα project έχουν επιλεγεί και ποιες είναι και, ποια είναι η εκτέλεση του προπολογισμού ε, ανά project. Μέχρι τώρα είχαμε κάποιες δυσκολίες με την εφαρμογή για διάφορους λόγους. Καταρχάς ε, υιοθετήθηκαν αργά κάποια προγράμματα. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι το ΕΤΘΑ είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα ταμεία γιατί είναι πιο συμπεριληπτικό. Έχουμε στήριξη για τις παραμεθόριες περιοχές, ε, για την θαλάσσια πολιτική. Ήταν αρκετά πιο περίπλοκο δηλαδή για τα κρατη να μπορέσουν να εκπονήσουν τα προγράμματά τους αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι καλύτερε τάσει ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Μα ε, είχαν ανησυχήσει αρκετά αυτά τα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα είναι η πρώτη χρονιά που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει και καθ' όλη τη διάρκεια τη προγραμματική περίοδου. Τώρα, ποια είναι κάποια από τα, ποιες είναι κάποιες από τις δραστηριότητε που α, ε, ε, χρηματοδοτούμε. Είπα ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά η ε, υποχρέωση εκφόρτωση είναι σημαντική. Ένας είναι αυτός από τους τομείς που έχουμε δεσμεύσει 88 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχουμε κάποια μέτρα όπως ο περιορισμός ε, του αντικτύπου στο θαλάσσιο περιβάλλον της αλίας, καινοτομία, προστιθέμενη αξία, ε, χώροι εκφόρτωσης, λιμένες και επίσης ανεπιθύμητα αλλιεύματα. Έχουμε 42 εκατομμύρια τα οποία έχουν δεσμευθεί για τις ε, προσωρινές παύσει, Όπως είπα πιο πριν, ε, εδώ μιλούμε κυρίως για κοινωνικο-οικονομικά μέτρα, τα οποία έχουμε για να επιτρέψουμε στους αλλοίς να ε, μπορέσουν να έχουν ένα ε, καλό επίπεδο διαβίωση όταν σταματά για οποιοδήποτε λόγο η λευτική του δραστηριότητα. α πούμε μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανανεώνεται. Οπότε αυτό σημαίνει μια ε, ανακούφιση για τον αλληλευτικό κλάδο ή κάποια βιολογικό, κάποιο είδου βιολογικού κλεισίματος. Ε, εκεί μπαίνει το μέτρο τη προσωρινή παύση. Έχουμε 96 εκατομμύρια ευρώ που πάνε στην μόνιμη παύση δραστηριοτήτων. Ε, για ε, ο παραπλησμός δηλαδή ε, των μόνιμων των, των αληφτικών σκαφών και αυτό γίνεται γιατί βεβαίω τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται το στόλο τους με τέτοιο τρόπο ώστε να πρέπει να προσαρμόσουν την ισορροπία μεταξύ της αλληλευτικής δυνατότητας και των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Οπότε μπορούμε έτσι μέσω αυτών των μέτρων να έχουμε πλήρη παραπλησμό των σκαφών. Επίσης, αντικατάσταση μηχανών δίνεται και εκεί κάποια χρηματοδότηση, εφόσον βεβαίω υπάρχει μείωση στην ισχύ τη μηχανή και εφόσον είναι πιστοποιημένε οι μηχανέ. Ε, η ισχύ, του δηλαδή. Θα έρθω λίγο αργότερα σε αυτό το θέμα όταν, μιλώ, όταν θα μιλήσω για την ε, μελλοντική πρόταση τη Κομισιόν. Έχουμε δαπανίσει αρκετά κονδύλια επίση στην ασφάλεια, την υγιεινή και τι συνθήκε εργασία. Μίλησα λοιπόν για κάποιου από του τομεί, ε, για τι αντιολιστικέ συμπογέ, για τι τουαλέτε, την ασφάλεια, τον εξοπλισμό, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν εμπίπτουν στο τρέχον ταμείο και θα συνεχίσουν να εμπίπτουν και να χρηματοδοτούνται και στο μελλοντικό ταμείο. Επίσης συνδράμουμε στο Natura 2000, έλεγχος και εφαρμογή, εκτέλεση έτσι και γενικώ διάφορα άλλα. Απλώς θέλω να έχετε μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε. Θέλω να τονίσω επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Φτάνουμε στις σε κάποιε από τι προθεσμίε για τους ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Θα έχετε ακούσει πολλή συζήτηση να γίνεται τι τελευταίε εβδομάδε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ή μάλλον η νέα πρόεδρο ε, θα ανακοίνωσε κάποιε νέε πρωτοβουλίε και τονίστηκε η σημασία του να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικέ μα θα ευθυγραμμιστούν με τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια των, ε, των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Έχουμε συγκεκριμένο στόχο για την αλληλεία, ο 14-6, που λέει και τον οποίο βεβαίω έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μέχρι το 2020 θα απαγορεύσουμε κάποια είδη ε, επιδοτήσεων αλληλεία που οδηγούν σε υπερδυνατότητα και υπεραλίευση και θα, απο... θα απορρίψουμε δυνατότητες που βοηθούν την υπεραλίευση και θα αποφύγουμε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. Ε, αυτή είναι η πρόταση που έκανε η Κομισιόν για το μελλοντικό ταμείο. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά. Σημαίνει ότι στο τρέχον ταμείο δεν έχουμε στήριξη για την κατασκευή, την αυπήγηση νέων σκαφών, κάτι που έρχεται από την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής του 2002, Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση εδώ και 20 χρόνια όπου τα δημόσια κονδύλια, τέλος πάντων τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια, δεν δαπανώνται για την ε, κατασκευή νέων σκαφών. Επίσης, δεν υποστηρίζουμε την αύξηση των ε, αλληλευτικών δυνατοτήτων. Το έτσα λοιπόν στην τρέχουσα μορφή του δεν επιτρέπει ε, οποιαδήποτε επένδυση που θα ενισχύσει την ε, αληφτική δυνατότητα και έχουμε και ειδικέ προποθέσει για τα μέτρα για τον στόλο. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε δαπανούμε, είτε για την κατάσταση μηχανή, είτε για την βοήθεια στου νέου αλληλεί να αρχίσουν την δική του επιχείρηση στον κλάδο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αποτρέψουν μια κατάσταση όπου πάλι θα έχουμε υπερβολικές δυνατότητες. Και θέλω εδώ πάλι να τονίσω το ότι το ΕΤΘΑ στην τρέχουσα μορφή του είναι λίγο το καμάρι των συζητήσεων που έχουμε με τις τρίτες χώρες, όπου λέμε ότι κοιτάξτε, είναι δυνατόν να υποστηρίξετε τον ελληνικό σας κλάδο σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, και τα οικονομικά μέτρα βιωσιμότητα, χωρί να δημιουργήσετε συνθήκε υπερβολική δυνατότητα ληφτική στον στόλο σα ή συνθήκε που θα οδηγήσουν σε υπεραλίευση. Αυτό ήθελα λοιπόν να το πω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, λίγα λεπτά ακόμη για την πρόταση του για το επόμενο ταμείο. Πολύ σύντομα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνδέσουμε τα όσα έχουμε στο τρέχον ταμείο με την νέα πρόταση που έχει υποβληθεί. Ε, να το δούμε ξεχωριστά, αν μου επιτρέπετε αυτό. Να ακούσουμε λίγο τα μέλη. Μας δώσατε κάποια γραφικά στοιχεία πριν. Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι για την εφαρμογή, για την εκτέλεση του προπολογισμού. Είπατε ότι έχουν ξεκινήσει τα πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και τώρα πάνε καλά. Αλλά εγώ έτσι όπως το ερμηνεύω το, το σημείο αυτό, ε, είπα, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είσαστε καθόλου κοντά στο να δαπανίσετε τα 6, τα δις που έχουν δεσμευθεί. Ένα από τα ε, σημεία κριτικής για το Ταμείο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να δαπανηθούν τα κονδύλια. Οπότε τι συμβαίνει πραγματικά και οι προβλέψει ποιε είναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει κάποια ε, χρήματα για να βοηθήσει τον ελληνικό κλάδο έτσι όπω προτείνεται. Αν δεν μπορούν να δαπανηθούν όμω τα χρήματα, εμεί δεν ε, τιμούμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει προ τον κλάδο. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Πράγματι είναι πολύ εύστοχη. Έχω να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, η τάση είναι πολύ πιο θετική από ό,τι υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Διαπιστώνεται δηλαδή επιτάχυνση ε, της ε, εφαρμογής. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα μέχρι το 2023 παρότι η προγραμματική περίοδος λήγει στο τέλος του 2020. Έχουμε το γνωστό κανόνα νη συν τρία ε, δημοσιονομικός κανόνας μεταξύ των πολλών που έχουμε. Αυτό, αυτός επιτρέπει ε, στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις δαπάνες των προγραμματικών ε, χρημάτων και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπάρχει δηλαδή μια περίοδος μετάβασης μεταξύ των δύο προγραμματικών περίοδων. Έχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη μέχρι το 2023. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση αφορά το Brexit. Εγώ ελπίζω να μην ε, επέλθει Brexit. Οι απώλειες και οι ζημίες ε, θα είναι για αμφότερες τις πλευρές της μάχης ε, τεράστιες και οι απώλειες αυτές φυσικά και οι ζημίες θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των τεράστιων ροών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και κατοχωρών. Αν ομιγέννητο γίνει ένα Brexit χωρίς συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές ε, όσον αφορά το κοινοτικό αλληλευτικό στόλο. Θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να δούμε πώς θα διατηρηθεί η αμοιβαιότητα και τα δικαιώματα πρόσβασης για τους αλληλείς μας ε, στα είδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του δικού μα αλείς στα νερά του Ηνωμένου Βασιλείου και του αλείς του Ηνωμένου Βασιλείου στα δικά μα. Οι ζημίε μπορεί να είναι τεράστιε. Παρατηρούμε ότι πολλά κονδύλια δεν έχουν δαπανηθεί και ήθελα να ρωτήσω στην εκπρόσωπο τη Κομισιόν, υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη ή αλλοί των οποίων αντιμετωπίζουν δυσκολίε λόγω του Brexit να μπορέσουν να λάβουν κάποια βοήθεια. Επίση, ήθελα να μάθω για πόσο καιρό μπορεί να προβλεφθεί μια τέτοια αποζημίωση. Δεύτερη ερώτηση, επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, διότι εδώ μα δείχνεται ότι 19,7% είναι το ποσοστό χρήση ε, του ταμείου. Δεν νομίζω να φτάσουμε στο 100% μέσα στα τρία επόμενα χρόνια. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος Οπότε τίθενται διάφορα ερωτηματικά. Πιστεύω ότι η κατάσταση δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η γραμματεία θα με επιπλήξει σίγουρα, αλλά γιατί πάντα κατηγορώ, καταγορώ τη γραμματεία, τον Κλάντιο εδώ, γιατί του αρέσουν οι ερωτήσεις της ομάδας για να επιταχύνουμε. Αλλά μια απάντηση, παρακαλώ, για αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση για την πρώτη ερώτηση του κ. Βαντάλεν έχω να πω δύο πράγματα. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν και τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα προσωρινής παύσης σε περίπτωση Brexit. Αυτή η πρόταση υιοθετήθηκε πριν μερικούς μήνες. Είναι έτοιμη. Αν επέλθει λοιπόν ε, αυτή η ανεπιθύμητη κατάσταση, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να αλλάξουν τα επιχειρησιακά του προγράμματα ανάλογα τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο που βλέπω με του συναδέλφου οι οποίοι εργάζονται στο επιχειρησιακό τμήμα βρίσκονται σε συνομιλίε με τα κράτη-μέλη που θα επηρεαστούν περισσότερο από το Brexit. Κάποια κράτη-μέλη ήδη τροποποιούν τα, τα επιχειρησιακά του προγράμματα για το ενδεχόμενο όπου αυτό θα συμβεί, ούτω ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και το Ταμείο να είναι έτοιμο να αποκριθεί. Όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, συμφωνώ μάλλον με τον κύριο Βαντάλεν. Είναι ανησυχητικό μεν, αλλά αν δει κανεί τι δαπάνε του δικού μα ταμείου σε σχέση με άλλα ταμεία, το κοινωνικό ταμείο για παράδειγμα, είμαστε λίγο πιο κάτω, αλλά περίπου στο ίδιο επίπεδο. Γύρω στα ίδια ποσοστά όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού είναι πιο αργό από ό,τι θα θέλαμε πράγματι, αλλά όχι τόσο δραματικό όσο τα περασμένα χρόνια. Παλιότερα ερχόμασταν εδώ στο Κοινοβούλιο, συζητούσαμε με τα κράτη-μέλη και τους λέγαμε παιδιά κοιτάξτε πρέπει να επιταχύνετε τις δαπάνε, πρέπει να ε, εντείνετε τις προσπάθειές σας, αλλά τώρα πραγματικά παρατηρούμε μία τάση ανωδική. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο σαφείς ε, όσον αφορά την απάντησή σας στην πρώτη μου ερώτηση. Επιτρέπετε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας για την αποζημίωση αλλιεών που θα έχουν ζημίες λόγω του Brexit και αν ναι, για πόσο καιρό. Εν συντομία, ναι είναι η απάντηση. Για εννέα μήνες. Και θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι στην απάντησή σας όσον αφορά την εκτέλεση. Πού βρέθηκε το πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στον ίδιο το μηχανισμό, ότι είναι πολύ γραφειοκρατικός, πολύ απλά, ή το πρόβλημα είναι τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν προτάσεις, ή ποιο, τι τέλος πάντων. Για ποιο λόγο είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όταν δίνουμε λεφτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν δίνεις απλά λεφτά. Είναι δύσκολη η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ξέρετε. Αν συζητήσετε με τους συναδέλφους που εργάζονται στη γεωργία, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στο κοινωνικό ταμείο, σε όλα αυτά τα ταμεία, υπάρχει κάποιος βαθμός πολυπλοκότητας διοικητικό άχθος. Γι' αυτό για την περίοδο μετά το 2020 έχουμε προτείνει σημαντικές απλουστεύσεις. η καθυστέρηση οφειλόταν σε κάποιο βαθμό στην καθυστερημένη υιοθέτηση κάποιων προγραμμάτων που υιοθετήθηκαν μερικά από αυτά τέλη του 2015, παρότι η προγραμματική περίοδος ξεκίνησε 1η Ιανουαρίου του 2014. Δεν θα κατηγορούσα λοιπόν τα κράτη-μέλη, ούτε μόνο την Κομισιόν και φυσικά όχι την Κομισιόν, εγώ προσωπικά όχι, αλλά είναι διάφοροι παράγοντε που εξηγούν το φαινόμενο αυτό, πρέπει να πω. Επίση, πρέπει να πούμε ότι ένα πράγμα που μα είπαν τα κράτη-μέλη είναι ότι ενίοτε όταν ανακοινώνουν προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ε, λαμβάνουν ελάχιστες αιτήσει. Δεν ξέρω αν επιλέγουν λάθος έργα ή δεν σχεδιάζουν τα σωστά έργα. Οπότε αυτό μπορεί να εξηγεί ε, τις καθυστερήσεις. Αν πάμε στην προγραμματική περίοδο 2007-2014 30% ε, του κονδυλίου του Ταμείου δεν δαπανήθηκε και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να μην ξανασυμβεί αυτό. Ένα τρίτο των χρημάτων δεν δαπανήθηκαν και χάθηκαν. Οπότε ελπίζουμε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στην τρέχουσα περίοδο. Μας βοηθήσατε πολύ με την απάντησή σας. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Sí, gracias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε κάποια πράγματα οι απόψεις μου δεν συμπίπτουν με την αξιολόγηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, ε, παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς την αιτιολόγησή του. Έχει δεν έχει καμία σχέση με το Ταμείο για τη Γεωργία, με το ΦΕΝΤΕΡ. Προγράμματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τις περιφέρειες. Εδώ μιλούμε για επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν σε ολόκληρα κράτη. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς αυτό, ναι, αλλά μετά να τηρήσει τις ε, ε, διατάξεις, τις περίπλοκες είναι εξαιρετικά επαχθές και δύσκολο. Δεν ξέρω Ποια είναι η πρόθεση της Επιτροπής. Είναι η πρόθεσή της να ταπανίσει, να σπαταλήσει χρήματα δεξιά και αριστερά. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει. Πρέπει να είναι κανείς πολύ δημιουργικός. Δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες για το πόσο γραφειοκρατικό άχθος συνεπάγεται το Ταμείο αυτό για το κλάδο. Και υπήρξε και μεγάλη καθυστέρηση στην έγκρισή του. Επομένως το 2019 πλέουμε με μια ταχύτητα η οποία οφείλεται μόνο στον άνεμο, χωρίς να στηρίζομαστε καθόλου σε μηχανές και κινητήρες. Άρα πλέουμε πάρα πολύ αργά. Μιλήσαμε για τις δαπάνες για τη μόνιμη την προσωρινή αναστολή, διακοπή. Η μόνιμη σταμάτησε πριν από κάποια χρόνια και συνεχίσαμε την προσωρινή για τα ε, βινθο είδη της Μεσογείου. Όταν δικαιολογείται ε, θα πρέπει να παραμένει αυτή η διακοπή, είτε μόνιμη είτε προσωρινή. Δηλαδή είναι πρόβλημα μεθοδολογίας. Και έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα να απευθύνω. Η εκπρόσωπος της Επιτροπή μίλησε για τα θέματα του ΦΙΛ και λέει το 14% των τοπικών ομάδων δράση, αυτοί που κάνουν τη διαφοροποίηση στις παράκτιες περιοχές, πρέπει να επενδυθεί σε θέματα φύλου. Δηλαδή το 14% πολύ λίγων χρημάτων το οποίο θα πηγαίνει στις ομάδες τοπικής δράσης πρέπει να κατευθυνθεί και στις υπόλοιπες πολιτικές καθόλου δεν θα υπάρξει η διάσταση του φίλου. Εκεί μόνο θα κάνουμε την προσπάθεια. Το είπε ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιήθηκε το 14% σε δράσεις των ομάδων ε, τοπικής δράσης για διαφοροποίηση κτλ. Σωστό, αλλά στις υπόλοιπες πολιτικές εκεί είναι ο μεγάλος όγκος. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για πράγματα του φύλου, για τη διάσταση του φύλου, γιατί είναι ευρωπαϊκό το θέμα. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Θέλω να πω το εξή μόνο. Επιτρέψτε μου. Τις τελευταίες ημέρες βλέπω ότι δεχόμαστε καταιγισμό mail, σπάμε ενδεχομένως, για τις υποτιθέμενες αυτοκτονίες στον αλλιευτικό κλάδο. Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Τη θέση αυτή την ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και την ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει είναι η εγκεκριμένη. Τη συζήτηση αυτή τη ζήτησαν κάποιες πολιτικές ομάδες. Πολύ ωραία να το συζητήσουμε και να συζητήσουμε και το μελλοντικό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά το Κοινοβούλιο τα έχει εγκρίνει αυτά κατά πλειοψηφία. Να μην δημιουργηθούν ψευδείς προσδοκίες και να μην νομίζουν ότι θα ξανακινήσει η συζήτηση. Ε, αυτό είναι αδύνατο εξ όσο γνωρίζω και θέλω να το διευκρινίσετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, να το ξεκαθαρίσετε γιατί υπάρχει διάφορος κόσμος που διαχειρίζεται και χειραγωγεί την κοινή γνώμη προσπαθώντας να ξανανοίξει το θέμα. Όμως στην προηγούμενη θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε απόφαση σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκάρσκιν, γιατί σίγουρα θα συμπληρώσει τα δικά σας λόγια κυρία Αγγιλέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας διηγηθώ λίγο τη ζωή μου και ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι από αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν το Ταμείο επί Επιτόπου. Ε, πριν από 7 χρόνια γινόμουν υποπεριφερειάρχης της περιφέρειας της Βρετάνης, ε, μια περιφέρεια η οποία αξιοποίησε ιδιαίτερο στο Ταμείο αυτό και θυμάμαι τη συζήτηση την έντονη εκείνη την εποχή και της παρουσιάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλεγε ότι θα δείτε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά. Λοιπόν, δεν είναι πιο απλά και δεν έγιναν πιο απλά. Ε, την απλούστευση δεν την είδαμε. Θα έπρεπε να είναι πιο απλά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Υπήρξαν καθυστερήσεις στην έγκριση, Είχαμε συζητήσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, συζητήσει με το Συμβούλιο. Λογικά είναι όλα αυτά, αναμενόμενα. Κάποιος χρόνος θα χρειαζόταν και χρειάστηκε. Όμως όταν ε, έγινε λόγος για την εφαρμογή του επιτόπου, εκεί υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις. Το αιώνιο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, επιβάλλει την περιπλοκότητα ή τα κράτη-μέλη ουσιαστικά υπονομεύουν τη δική τους την πορεία. Δηλαδή ένας αλλιέας θέλει να ζητήσει επιδότηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Πηγαίνει στο διαδίκτυο. Πρέπει να το εκτυπώσει 50 σελίδες. Έστω το εκτυπώνει. Συνήθως πάει σε μια συμβουλευτική υπηρεσία, σε ένα εξωτερικό γραφείο που το βοηθά να συμπληρώσει και με το χέρι συμπληρώνει τις πέντε σελίδες, μια δουλειά πολύ μακροσκελής, βάζει τρεις προσφορές για κάθε μια πιθανή δαπάνη, τα βάζει σε ένα φάκελο, τα στέλνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου ε, τα ανοίγουν όλα αυτά, τα σκανάρουν και μπαίνουν στον υπολογιστή τους και με το πληκτρολόγιο περί... Ε, βάζουν στον υπολογιστή το περιεχόμενο. 8 ώρες δουλειά για έναν υπάλληλο της περιφέρειας. Δηλαδή, εδώ σταματώ καταρχάς για να πω ότι θα μπορούσε ο Αλιέας ή το συμβουλευτικό του γραφείο να τα συμπληρώσει όλα αυτά διαδικτυακά. Το ίδιο θα ήταν. Αυτά για την ολοκλήρωση του φακέλου. Μετά, για την πληρωμή δύο φορές από 8 ώρες για τα στελέχη της περιφέρειας, χίλιοι φάκελοι του Ταμείου για την περιφέρεια της ε, Βρετάνης, ε, δηλαδή ένα πλήρες ωράριο των στελεχών του Δημοσίου 2.000 ημέρες. 10 θέσεις απασχόλησης το χρόνο. Φτάνει μια στιγμή λοιπόν που λέει κανείς η Γαλλία τα έχει κάνει αυτά, τα γραφειοκρατικά κτλ. Ε, έτσι ήταν όμως. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σημειώνονται καθυστερήσεις και έχουν σημειωθεί τόσες πολλές καθυστερήσεις που μετά υποχρεωνόμαστε να λέμε ότι πρέπει να τα ξοδέψουμε για να μην χαθούν τα κεονδύλια, να τα, να τα ξοδέψουμε, να τα ξοδέψουμε. Και άρα χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο τη στρατηγική προσέγγιση. Τα δεχόμαστε ό,τι μας φέρνουν και ό,τι μας σερβίρουν το δεχόμαστε για να υπάρξουν τα πάντα και απορρόφηση κονδυλίων. Τώρα αν αυτά δώσουν κάτι και αποφέρουν κάτι ουσιώδες, αυτό είναι μαχητό και δεν τεκμέρεται δείξατε τα νούμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, με τις δεσμευμένες πιστώσεις και με τις δαπανηθήσεις πιστώσεις. Όμως, υποτίθεται ότι το Ταμείο πριν από 7 χρόνια μας είπαν ότι θα ήταν προσανατολισμένο προς τα αποτελέσματα και όχι προς τις δαπάνες. Ποια είναι λοιπόν τα αποτελέσματα, τα απτά αποτελέσματα. Αυτό ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόλερ, ακούσαμε δύο ερωτήσεις για την περιπλοκότητα του μηχανισμού και ξέρω ότι αναζητείτε λύσεις, αλλά ε, είναι τέσσερα χρόνια μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα. Γιατί δεν μπορούν να απλουστευτούν τώρα τα πράγματα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε τέσσερα χρόνια. Αυτή η Επιτροπή φταίνε τα κράτη. Πείτε μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Καλίνσκι τα συνόψισε πολύ σωστά όταν είπε ότι τίθεται το αιώνιο ερώτημα. Οι κανόνες φταίνε ή ο τρόπος με τους οποίους εφαρμόζουν, τους εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Και εγώ ε, σχόλια σε αυτό το θέμα την πρώτη φορά που πήρα το λόγο. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πολλών και διαφορετικών πραγμάτων. Πράγματι, σε επίπεδο κράτους ενίοτε υπάρχει αυτή η έννοια της ε, αστραφτερής πινακίδας. Δηλαδή έχουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και προστίθενται εθνικοί και τοπικοί έτσι ώστε να έχουμε ένα οικοδόμημα περίλαμπρο ε, που να λάμπει. Από μέσα όμως υπάρχουν καθυστερήσει, παρεμποδίζονται τα πράγματα από το να προχωρήσουν γρήγορα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε θέματα απλούστευση. Πλησιάζουμε προ το τέλο τη προγραμματική περίοδου. Ήταν όμω βασική μα περίγη έμπνευση για την πρότασή μας για το μέλλον. Τα έχουμε απλουστεύσει για το, μελά, για το μετά. Δεν θα έχουμε προγραμματισμό με βάση ε, τα μέτρα θα έχουμε προτεραιότητες στην πρότασή μας για το μετά και θα τα εξηγήσω αργότερα όλα αυτά. Τώρα, η κυρία Αγγιλέρα έχει δίκιο. Ο αφοπλισμός των αλληλευτικών σκαπών, το να πάνε για παλιοσίδερα, είναι κάτι που χρηματοδοτείται από το Ταμείο μέχρι τα τέλη του 2017. Έγινε όμως εσκεμμένα η επιλογή των συνομοθετών. Υπάρχει σταδιακή εξάλληψη, δηλαδή με τη μεταρρύθμιση του 2013 το Ταμείο θα έπρεπε να δείξει, να αναπαραστήσει την φιλοδοξία αυτής της μεταρρύθμισης του 2013. Και τώρα έχουμε επανεισάγει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το Ταμείο για να επιδοτηθεί ο αφοπλισμός και η απόσυρση των αλευτικών σκαφών και για την περίοδο μετά το 2020, γιατί πράγματι εξελίξεται η κατάσταση και πρέπει το Ταμείο να είναι αρκετά ευέλικτο για να αντιαποκριθεί και σε αυτές τις προκλήσεις. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημά σας για το φύλλο και τη διάσταση του φύλου. Το στατιστικό στοιχείο του 14% που έδειξα το έκανα για να δείξω ότι όλα τα project, όλα τα έργα που ενισχύονται, που επιδοτούνται με κοινοτικά και κονδύλια σε τοπικό επίπεδο έχουν συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου κατά 14% σίγουρα και αφορούν ε, και τον τομέα της αλίας και άλλες παράκτιες κοινότητες. Δεν είναι τα μόνα έργα του ταμείου που έχουν διάσταση του φύλου ε, σωματωμένη. Για παράδειγμα, στην υδατοκαλλιέργεια χρηματοδοτούμε διάφορες start-up, τις οποίες έχουν γυναίκες. Έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που συχνά ε, έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση των γυναικών στο σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν στον κλάδο της αλληλείας. Θέλω αυτά να τα διευκρινίσω λοιπόν. Τώρα, για το ερώτημα του κύριου Καρλίνσκι, ποια είναι τα αποτελέσματα. Προσπάθησα στην παρουσίασή μου κάποια να τα εξηγήσω. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το στάδιο. Τώρα φτάνουμε στην ταχύτητα πλεύση στην κανονική, σε μια κανονικότητα δηλαδή, οπότε είναι νωρίς να μιλήσουμε για αποτελέσματα, αλλά σας έδειξα ήδη ένα παράδειγμα. Το 14% όλων των έργων έχουν στόχο τις γυναίκες. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό. Έχουμε δει μείωση στη συνολική δυναμικότητα του στόλου. Και αυτό είναι θετικό και είναι χάρη στα χρήματα που δίνουμε για τον αφοπλισμό, για την απόσυρση δηλαδή, για τον παροπλισμό μάλλον, όχι αφοπλισμό, ζητά συγγνώμη δερμηνέας. Και πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν κέρδη 1,3 δις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο της αλληλείας. Πόσα από αυτά είναι και χάρη στο Ταμείο, ε, αυτό είναι αυτό που θα μας απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και αξιολογητές οι ειδικοί. Έχουμε όμως άποψη από αυτού. Και θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ πιο κερδοφόρα, ε, κερδοφόρα περίοδος από ό,τι στο παρελθόν και χάρη στην βοήθεια του Ταμείου. Εγώ πιστεύω ότι το Ταμείο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Ε, σταματώ κάπου εδώ. Ελπίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος των ομιλητών. Να μην ξεπεράσει τα δύο λεπτά ο καθένας, παρακαλώ, γιατί... Ε, δεν θέλω να έχουμε πολλές ομαδικές ερωτήσεις, γιατί όσο περισσότερο τις γκρουπάρουμε τις ερωτήσεις, τόσο πιο γενικές είναι οι απαντήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι διότι επιταχύνεται ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων. Η καθυστερημένη έγκριση του προγράμματος ήταν ένας από τους βασικούς λόγους καθυστέρησης, άλλωστε το λένε και οι εμπειρογνώμονες. Πρέπει να γίνει ένα ταμείο πιο εύκολο προς τη χρήση του, γιατί είναι περίπλοκο αυτή τη στιγμή και ούτω καθεξής. Έχω τρία ερωτήματα να απευθύνω. Ποιος είναι ο αριθμός των αλλιευτικών σκαφών που έχουν οφειληθεί από το Ταμείο και σε ποιο ποσοστό το έχουν χρησιμοποιήσει σκάφη που προέρχονται από την ερεστεχνική αλία, την, την αλία μικρής κλίμακας. Έχετε νούμερα και ποσοστά για αυτές τις αναλογίες. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Τα περιβόητα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να περιλαμβάνονται και στο νέο ταμείο σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήθηκαν. Μέρος των ενισχύσεων σε ποιο βαθμό συνοδεύτηκαν από ε, ε, τέτοιου είδους εργαλεία. Έχετε περισσότερα στοιχεία και πιο ακριβή κυρίως. Και τρίτο ερώτημα για τον εξυγχρονισμό των κινητήρων των αλληλευτικών σκαφών. Ε, η αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο ήταν πολύ περιορισμένη. Έχετε στοιχεία γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόλερ, έχετε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις τεκμηριωμένες. Είστε σε θέση να δώσετε σαφείς και ακριβείς απαντήσεις. Έχω και διαφάνεια. Περιμένετε να τη δείτε. Κρατηθείτε. Πού είναι η διαφάνειά μου. Έρχεται. Λοιπόν, θα χρησιμοποιούσα αυτή τη διαφάνεια στην επόμενη μου παρουσίαση, αλλά ο κύριος Μιγιανμόν ρώτησε πόσα αλληλευτικά σκάφη ωφελούνται από το Ταμείο. Δεν έχω το ακριβές νούμερο. Όμως, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε περίπου 10.000 έργα. Το 52% του Ταμείου έχει στραφεί προς σκάφη αλίας μεγάλης κλίμακας. 7.500 project για την αλία μικρής κλίμακας, άρα το 41% των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ταμείο μας αφορούν σε σκάφη αλίας μικρής κλίμακας. Αυτό σε νούμερα μεταφράζεται ως εξή. 70% της συνολικής χρηματοδότησης πηγαίνει στη μεγάλη κλίμακας και 18% στην αλία μικρής κλίμακας. Αυτό βεβαίως δεν αντιπροσωπεύει αναγκαστικά τον αριθμό των μεγάλων και των μικρών αλλιευτικών σκαφών που έχουμε, γιατί το 75% του στόλου είναι μικρής κλίμακας. Άρα, δυστυχώς, το Ταμείο δεν ε, ε, ευνοεί το σύνολο του κλάδου και τίνει να ευνοεί τον, τον, τον στόλο μεγάλης κλίμακας που ουσιαστικά είναι μόνο το 20% του στόλου συνολικά. Τώρα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ένα κράτο μέλο στην Εσθονία που αξιοποιεί τέτοιου είδου χρηματοδοτικά εργαλεία στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Τη Δευτέρα είχα μια συζήτηση με τα κρατη και υπάρχουν και άλλα από ό,τι φαίνεται που θα θέλουν να αξιοποιήσουν τέτοιου είδου χρηματοδοτικά ή οικονομικά εργαλεία. Έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων, η οποία προσφέρει στήριξη σε κράτη που θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιου είδου χρηματοδοτικά εργαλεία, δάνεια με εγγυήσει, με το κ.ο.κ. Και για την αντικατάσταση των κινητήρων. Πράγματι, δεν έχει αξιοποιηθεί ιδιαίτερο σε αυτό το μέτρο. Θα έλεγα ότι χίλιοι κινητήρε έχουν αντικατασταθεί. Αυτό όμως οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι Έχουμε την υποχρεωτική απέτηση μείωση τη υποδύναμης του κινητήρα και ίσως αυτό δεν είναι και τόσο ελκυστικό ω επιλογή για τον κλάδο, να υποβάλει έτοιμα δηλαδή για να ενισχυθεί, να δεχθεί ενίσχυση και επιδότηση για να αντικαταστήσει κινητήρα με κινητήρα μικρότερης υποδύναμης. Ελπίζω ότι απάντησα σε όλα σα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριο Σαλάκ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω Γάλλος που εκπροσωπώ την Σκοτία η Μεγάλη Βρετανία είναι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσει να είναι. Ε, να πω στον κύριο Βαντάλεν, είπε ε, πολύ σωστά ότι το Brexit ε, είναι μια κατάσταση όπου χάνουν όλοι. Έτσι έχει, αν δει κανεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, το οποίο θα πάψει να βοηθά το Ενωμένο Βασίλειο. Το Ενωμένο Βασίλειο τα πήγαινε πολύ καλά και ειδικότερα η Σκωτία. Αν δείτε τα νούμερα μέχρι στιγμής φέτος, το τελευταίο γύρο που τελείωσε 30 Σεπτεμβρίου μπορώ να σας πω επίσημα ότι η χρηματοδότηση υπήρξε άνευ προηγουμένου. Και τώρα χρειάζεται να κλείσουμε τις νέες εφαρμογές για πολλά από τα μέτρα, διότι δαπανίσαμε όλα τα χρήματα που μας συγχωρήθηκαν. Αυτά είναι καταπληκτικά νέα. Είναι δηλαδή εφικτό τα καταφέραμε εμεί και θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε παράδειγμα και για άλλου. Μπορώ να σα πω για παράδειγμα ε, δύο εργοστάσια επεξεργασίας ε, ε, αλλιευμάτων 100 μέτρα από εκεί που ζω στο Αμπερντίν κέρδισαν, ε, έλαβαν πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες ε, λίρες από το IMF, e ε, κάτι που θα χαθεί τώρα, αλλά όπως είπα το Brexit δεν θα συμβεί, οι περισσότεροι είμαστε εδώ, τα περισσότεροι αιρετοί του Ηνωμένου Βασιλείου είπαν δεν θέλουν το Brexit, είμαστε πλειοψηφία και εδώ και σε αυτή την Επιτροπή και λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνει το Brexit, τα δικαστήρια συμφωνούν μαζί μας, οπότε θεωρούμε ότι το μέλλον διαγράφεται θετικό. Έχω μία ερώτηση. Αφού η Σκοτία τα πάει τόσο καλά στις δαπάνες, τι είναι αυτό που κάνει σωστά και τι κάνουν λάθος οι άλλε χώρε, τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Και αν τα άλλα κράτη δεν μπορούν, μήπως να δαπανίσουμε όλα τα χρήματα στη Σκωτία. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχει τρόπο. Θα μα άρεσε όλου. Καταπληκτικά που η Σκοτία ξοδεύει τα χρήματα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια άλλη έκθεση όπου τα χρήματα των φορολογουμένων πάνε να επιδοτούν απαράδεκτες δραστηριότητες όπου μου είπαν την περασμένη εβδομάδα να ασχολούμαι με τα δικά μου προβλήματα. Ένας Γάλλος ε, βουλευτή που δεν του άρεσε αυτά που είπα εγώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καταλάβει ξανά ε, τις θάλασσές της. Να είχατε δώσει τις ίδιες ε, συμβουλές όταν το, δόθηκε το τελεσίγραφο ε, στη Ηνωμένο Βασίλειο. Για μένα τέτοιου είδους συμπεριφορά θα ανάψει τα πνεύματα, εκτός αν βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε τον Brexit. Όπως είπε ο κύριος Βαντάλεν, χρειαζόμαστε έναν καλύτερο τρόπο. Ο θυμό και οι απειλέ για τα Ιναλία έχει ξεκινήσει ήδη και η Βρετανία δεν έχει ακόμα αναχωρήσει. Δεν νομίζω ότι κανείς μας εδώ που να υποστηρίζει το Brexit ή όχι θέλει να επαναληφθεί η μαγιά των Γάλλων που είδαμε πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός πρέπει να συμβιώσουμε, να συνεργαστούμε και να έχουμε και εμπορικές συναλλαγές. My turn. For... Excuse me. For 40 years... Για 40 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράζεται τα αλλιεύματα του και παρέχει ε, πολύ, καλή, ε, ε, πολύ καλά εισοδήματα σε ξένους αλληλείς Αλλά αυτές οι μέρες τελειώνουν όπως ένα διαζύγιο το Ηνωμένο Βασίλειο ξαναπαίρνει αυτό που είχε φέρει στο γάμο και απαιτεί να ξαναγίνουν δικά του τα υδατά του και αντίθετα με οποιοδήποτε διαζύγιο πρέπει να αποδεχθείτε την κατάσταση για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σταματήσετε τη ρητορική και να αρχίσετε να δέχεστε ότι θα γίνει το Brexit. Ευχαριστώ φίλοι μου. <laughs> Δεν νομίζω ότι η κυρία Λάρντ ρώτησε κάτι. Ε, να προσπαθήσουμε παρακαλώ οι επόμενοι να μείνουμε και εντός των χρονικών ωρίων. Ο κύριος Ρόιτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγο να επανέλθω σε αυτό που συζητούσαμε πριν ε, κάνουμε αυτή την ε, αλλαγή ρότας προς τον Brexit. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικά τα όσα ακούσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ε, υπάρχει, υπήρξε αργή έγκριση του προγράμματος και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ουσιαστικοί λόγοι που έγινε αυτό για τη χρήση των κονδυλίων. Εντάξει, μερικώς αυτό μπορεί να οφείλεται και στους περίπλοκους κανονισμούς και στο διοικητικό άχθος, στη γραφειοκρατία. Αλλά αν δούμε και τη διαφάνεια, Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ε, υπάρχει η ίδια κατάσταση για την χρηματοδότηση. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν πιο υψηλέ ε, αιτήσει. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν πολύ χαμηλά στατιστικά. Ε, η Κομισιόν έρχεται σε επαφή με τα κράτη-μέλη, τους μιλάει, προσπαθεί να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν. Μιλάτε με τα κράτη-μέλη για τις βέλτιστες πρακτικές, ας πούμε, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα ενθαρρύνετε να υποβάλουν περισσότερε αιτήσει και να λάβουμε περισσότερα κονδύλια. Νομίζω ότι είναι μεικτή ευθύνη εδώ. Και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη και η Κομισιόν. Η Κομισιόν λοιπόν από τη δική τη τη μεριά τι κάνει για να μπορέσει να πιέσει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν περισσότερε αιτήσει. Και για τον Brexit πρέπει να πω ότι. Ε, εντάξει να έχουμε ελεύθερο εμπόριο, αλλά η πρόσβαση στα ύδατα ημέν των άλλων είναι πολύ περίπλοκο θέμα και σίγουρα θα είναι πολύ περίπλοκες και αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει. Ναι, Πρόεδρε, για την χαμηλή εκτέλεση. Αν ήμουν εδώ πέρσι, θα σας έλεγα ότι ανησυχώ. Φέτος δεν ανησυχώ τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί αν δείτε συνολικά τα στατιστικά για το ευρωπαϊκό ε, οικοδόμημα, είμαστε στο 44% των ε, επιλογών επιχειρήσεων. Είμαστε στο τέλος του 2019 σχεδόν, άρα έχουμε τέσσερα ολόκληρα χρόνια δαπανών διαθέσιμων δαπανών. Οπότε εγώ δεν ανησυχώ όσο ανησυχούσα πέρσι. Αν καθόμουν εδώ πέρσι θα σας έλεγα ναι, είναι πολύ δύσκολο, είναι περίπλοκο, ανησυχούμε, αλλά φέτος δεν ανησυχούμε τόσο πολύ. Αυτό που κάνουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη όπου έχουν χαμηλή εκτέλεση, είναι ότι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα των, επιχειρησιακών ε, ε, δραστηριοτήτων έρχονται σε επαφή με, τις, με τα κρατημέλη, συμμετέχουν στις ε, προπαρασκευαστικέ ε, συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις της αναθεώρησης, όπου ε, κάνουμε αναπροτεραιότητα συζήτηση για το πού είναι τα προβλήματα και πού υπάρχουν δυνατότητες καλύτερης εκτέλεσης. Μία από τις δυνατότητες των κρατών μελών, και το κάνουν φέτος, είναι να μετακινούν κονδύλια από τις χαμηλής δαπάνης προτεραιότητας στις υψηλής δαπάνης. Και αυτό γίνεται και στα πλαίσια τη αναθεώρηση των επιδόσεων που γίνεται και φέτο. Πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει αυτή τη μεταφορά, έχουν τροποποιήσει τα επιχειρησιακά του προγράμματα και μπορούν να μετακυλίουν τα κονδύλια από τι χαμηλέ προτεραιότητε στι υψηλέ. Και αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο. Σύντομα. Ελπίζω να απήντησα σε όλε τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμάτου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι το επίπεδο των πληρωμών όσο οι δεσμεύσεις για να λείψει υποχρεώσεων. Ε, ε, υπάρχει ο κανόνας νήσιν 3, πράγματι. Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στην νήσιν 2, όπως προτείνεται για τα διαρθρωτικά ταμεία, για το κοινωνικό ταμείο, για παράδειγμα. Διότι αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι οι διοικήσει μας, και εδώ είναι αυτό καταγγελία αυτό που λέω, ξένε ότι είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε, οπότε επιταχύνοντας επηρεάζεται η ποιότητα της δαπάνης και προσωπικά γνωρίζω υποθέσεις περιφερειών που δαπανούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δυστυχώς για την ανανέωση του αστικού τοπίου για παράδειγμα σε μέρη τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα σίγουρα αλλά δεν αποτελούν πραγματικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Ελίας εκεί χάνονται τα χρήματα αντιθέτως οι Ελίες μας ξαφνικά υποχρεώνονται να βάλουν ε, λεφτά από την τσέπη τους στη συγχρηματοδότηση. Οπότε αυτό που με ανησυχεί ε, είναι, είναι, έχει λογική καλύτερα να επιστρέψουμε στο νησιν και καλύτερα έλεγχη μήπως θα ήταν προτιμότερη. Ευχαριστώ. Um, Mrs. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσία της εδώ. Δεν θα μπω στην περιπλοκότητα του εγχειρήματο και στην αδύρυτη ανάγκη απλούστευσης του. Έχω όμως ένα ερώτημα να θέσω στην Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την αξιοποίηση των πόρων με μεγαλύτερη αποκέντρωση. Το πιστεύει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια να εφαρμόσουμε τη διάσταση της περιφέρειας. Είναι κάτι που έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερο στη νέα μεταρρύθμιση της αλλιευτικής ε, πολιτικής. Είναι μια δυνατότητα αυτή η αποκέντρωση για το πώς χρησιμοποιούνται τα προγράμματα από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, έχετε νούμερα για το αριθμό των σκαφών που προχωρούν σε εκφορτώσεις. Πόσοι ε, που προχωρούν σε παραπλησμό. Πόση είναι η μείωση της απασχόλησης λόγω των σκαφών που παροπλίζονται; Έχετε νούμερα για τις νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια ή δεν δημιουργήθηκαν. Τώρα για τη μείωση του αριθμού του στόλου μετά από σημαντική μείωση, τουλάχιστον σε ορισμένε περιφέρειε και σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η τραγική μείωση σκαφών είναι συμβατή με την απέτηση εξυγχρονισμού η οποία συνοδεύεται και εξυγχρονισμό με την, της υποδύναμης. Δηλαδή η υποδύναμη του κινητήρα είναι αυτή η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια του σκάφους όταν βγαίνει να αλλιεύσει στην ανοιχτή θάλασσα. Και για το θέμα του Brexit και της Σκοτίας, ε, βέβαια δεν με αφορά εμένα, θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση. Α, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τα δικαιώματα τα αλλιευτικά που έχει, πόσα είναι της Σκοτίας. Αυτή η απάντηση μπορεί να μας δοθεί για να μπορώ να φανταστώ κι εγώ υποθετικά μελλοντικά σενάρια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν κύριο θα ακούσουμε πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω ως φιλελεύθερος σήμερα. Οικονομικά φιλελεύθερος ενώ που συχαίνεται τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις στρεβλώνουν την κατανομή των πόρων. Απομακρύνουν από την παραγωγική χρήση στη μη παραγωγική το ότι ένα, το προηγούμενο ταμείο είχε 30% ε, που δεν δαπανήθηκε δείχνει την αποτυχία του κεντρικού προγραμματισμού. Οι επιδοτήσεις ε, ανταμείβουν τους παραγωγούς εις βάρος των καταναλωτών. Σε αυτή την περίπτωση εις βάρος της ε, αλληλευτικής βιωσιμότητας. Το να επιδοτούμε την κατασκευή αλληλευτικών σκαφών όταν ανησυχούμε για τη διατήρηση των ψαριών είναι τρέλα είναι σαν να ρίχνεις πετρέλαιο πάνω σε μια φωτιά. Ο κύριος Βανταλέν ρωτά αν τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις, αυτά που δεν πανήθηκαν. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί να μην τα επιστρέψουμε στους φορολογούμενους. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό με εκπτώσεις ε, στις ε, ε, χώρες που συμβάλλουν και ρωτώ την Επιτροπή έχετε επιστρέψει τα χρήματα σε αυτούς που τα έδωσαν. Ναι. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις ακόμα, αλλά θέλετε να απαντήσετε στα γρήγορα σε αυτά που μόλις ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το νησιν 2 ή νησιν 3. Στην πρόταση της Κομισιόν για, μετά το 2020 για όλα τα ταμεία έχουμε προτείνει να επιστρέψουμε στο νησιν 2 και όχι στο νησιν 3. Γιατί? Τα νούμερα πιστεύω που μόλις σας έδειξα δείχνουν το γιατί. Το πρόβλημα είναι ότι αν επιλέξεις τον ΙΣΙΝ 3 δεν υπάρχει κίνητρο στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν αρκετά γρήγορα τα προγράμματά τους και να αρχίσουν να δαπανούν. Απλά παρατείνησε την ημερομηνία λήξη του προγράμματο. Για αυτό του λόγου, μεταξύ άλλων, η Κομισιόν προτείνει να επανεισαγωγεί του νησιν Η δεύτερη ερώτηση αφορά την αποκέντρωση το ακούσαμε από πολλούς προλαλήσαντες γιατί δεν έχουμε περιφερειακά προγράμματα στο EMFF διότι είναι πολύ μικρό, πολύ απλά. Ας δούμε την υπόθεση της Γερμανίας. Ε, την περίπτωση της Γερμανίας που είναι ένα αποκεντρωμένο κράτος ε, με πολλές αρμοδιότητες για τα, για τα κρατήδια. 260 εκατομμύρια εκχωρούνται σε αυτή την περίοδο για τη Γερμανία δια 7 έτη, δια ε, τον αριθμό των κρατηδίων δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό. Δεν έχει νόημα να έχουμε ένα περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο λόγος. Για την ε, καταστροφή πλοίων δεν έχω αρκετό νούμερα για το πόσα πλοία διαλύθηκαν αλλά δαπανίσαμε 96 εκατομμύρια για τη διάλυση πλοίων στην τελευταία περίοδο. Είναι πολλά πλοία δηλαδή. Τώρα, για αυτό που ανέφερε η κυρία Μπιλμπάου, η συνοχή μεταξύ του να ε, ζητάς διάλυση ή ε, θέση εκτός λειτουργίας με δημόσια χρήματα ε, για σκάφη και να ζητάς εξυγχρονισμό και αναβάθμιση και κατασκευή νέων σκαφών. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε ένα πράγμα. Αν δεν δείχνουμε συνοχή στα όσα λέμε, λέγοντας ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο για να διαλύσουμε πλοία και για να κατασκευάσουμε νέα, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει από άψη συνοχή. Η τελευταία ερώτηση που θέλω να απαντήσω για τα χρήματα που δεν έχουν δαπανηθεί, ο κανόνας νήσιν 3 λέει ότι οποιαδήποτε χρήματα δεν δαπανηθούν επιστρέφουν στον προϋπολογισμό και τελικά στα κράτη-μέλη. Τα χρήματα δηλαδή τελικά επιστρέφονται στο κράτος μέλος που τα έδωσε τα μη δαπανηθέντα κονδύλια, δηλαδή δεν ανακατανέμονται σε άλλου τομεί. Αυτό ελπίζω να απάντησα σε όλε τι ερωτήσει. Ο κ. Μωτήθ είναι ικανοποιημένο. Ε, ε, πιο ικανοποιημένο, λέει ο κ. Μωτήθ. Λοιπόν, τελευταίο γύρο έχουμε τρει ομιλητέ. Κλείνω τον κατάλογο. Κυρία Μοντέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις. Παρά τις εξελίξεις, τις οποίες ξέρουμε, το ΕΤΘΑ είναι ένα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, την ε, χαμηλότερο, με το χαμηλότερο ρυθμό δαπανών, που κατά συνέπεια θα οδηγήσει το Συμβούλιο να αλλάξει λίγο την κατάσταση και να μην επιτρέψει να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις στο Ταμείο. σε ό,τι αφορά την ανανέωση των γενεών και τα λοιπά, τα περιβαλλοντικά μέτρα αυτό και την βιώσιμη, βιωσιμότητα μπορεί αυτό να λειτουργήσει καλά. Αλλά όταν μιλούμε ας για την στήριξη για τα σκάφη, ε, πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και εννέα υπερπεριφερειακές ε, ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν αλληλεία μικρής κλίμακος και μια παράδοση αλίας μικρή κλίμακος και τα σκάφη είναι πολύ μικρότερα από αυτά που χρησιμοποιούνται από στόλου άλλων περιοχών της Ευρώπης. Μόλι το 19% των κονδυλίων ε, αποδίδεται στη στήριξη τέτοιου είδου μικρών σκαφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει τα, τελευταία, τα επόμενα συγγνώμη, τέσσερα χρόνια και για να μειώσει τη γραφειοκρατία και για να δώσει στήριξη σε αυτά τα είδη ε, σκαφών και σε αυτού του αλληλεί οι οποίοι βεβαίως βρίσκονται εκεί υπό πολύ μεγαλύτερη πίεση. Το άρθρο 249 τονίζει τη σημασία αυτών των υπερπεριφερειακών ε, περιοχών, οπότε εσείς τι μπορείτε να κάνετε με ένα θετικό πρόσημο για να μπορέσετε να βοηθήσετε και να προστατεύσετε αυτά τα σκάφη και αυτού του αλληλείς, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να συνεχίσουν να αλλιεύουν και να, ε, βελτιώ... να αλλιεύουν με καλύτερο και βιώσιμο τρόπο. Θέλετε να του ε, βοηθήσετε, όλοι θέλουμε να του βοηθήσουμε δηλαδή σε αυτές τις ε, περιοχές, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στα δικά τους χαρακτηριστικά. Οπότε τα επόμενα χρόνια εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθηθούν ε, αυτή η ελίς. Πώς μπορεί αυτό το 19% να βοηθήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αρκετό για να βοηθήσει τέτοιου είδους ε, αλείς. Έχω κάποια αιτήματα ακόμη για ε, παρεμβάσεις, αλλά επειδή και το επόμενο σημείο για το ΕΤ θα είναι, για το επόμενο πρόγραμμα, φαντάζομαι θα μπορέσετε να, βάλετε την, να θέσετε τη συζήτησή σας σε εκείνο το σημείο. Κυρία, Σάλιβαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν χώρες που είναι καλές στην απορρόφηση κονδυλίων. Υπάρχουν χώρες που είναι κακές στην απορρόφηση κονδυλίων και η Κομισιόν τι κάνει σχετικά για να υποστηρίξει τις χώρες που δεν τα πάνε και τόσο καλά σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων. Και σε σχέση το, το, το, με τα όσα είπε ο κύριο Σάλλαρντ για τη Σκοτία, που είναι τόσο επιτυχής και το και μπορεί να στηρίξει καλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα σαν τη σκοτία χωρών που εποφελούνται όντως από το κονδύλιο του Ταμείου και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υποδείγματα για άλλες χώρες. Καλή ερώτηση. Κύριε Κόμπερτ, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Πρώτη για το θέμα αυτό το περίφημο των επιδοτήσεων για την κατασκευή. Και στις, ε, στην προηγούμενη θητεία πριν τις εκλογές είχαμε ψηφίσει υπέρ. Αυτό μπορεί πλέον να μην είναι θέση του νέου α, κοινοβουλίου γιατί είχαμε, τέλει, έχουμε πια διαφορετική σύνθεση του κοινοβουλίου οπότε βεβαίω το ερώτημα δεν είναι για εσά, πρόεδρε αλλά τι δυνατότητε έχουμε να ξανααναθεωρήσουμε μάλλον αυτή τη θέση και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποσύρει την υπάρχουσα πρόταση. Βεβαίω, πάντα μπορεί να αποσύρει προτάσει η Κομισιόν, αλλά μπορεί να, υποβάλει, να ξανά υποβάλει αυτή την πρόταση, έτσι ώστε να, να, να πιέσει με κάποιο τρόπο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσουν τι απόψει του σε σχέση με κάποια στοιχεία τη πρότασή του. Δεύτερο ερώτημα. Ε, θαλάσσια απόβλητα. Τα ξέρουμε όλοι τα προβλήματα των α, αλλιέων που πρέπει να συλλέγουν τα, α, τα απορρίμματα και καμιά φορά όταν α, ε, έφερναν, τα έφερναν τα απορρίμματα πίσω, τα απόβλητα πίσω στο λιμάνι, έπρεπε να πληρώσουν και πρόστιμο. Του ε, κατηγορούσαμε κιόλα. Μερικώς ε, το ΕΤ θα έχει κάποια κίνητρα για να ενθαρρύνει τους αλληλείς να συλλέγουν τα απόβλητα, τα θαλάσσια, αντί να τους ποινικοποιεί. Ε, και επίσης, αν κατάλαβα καλά, η απορρόφηση ήταν πολύ χαμηλή σε αυτό το τομέα. Ε, φαντάζεστε ότι θα αυξηθεί, θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ε, μπήκατε κατευθείαν στα χωράφια του επόμενου σημείου, κύριε Κόμπερτ. Αν, ε, επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα, θέλω να σα θέσω κι εγώ ένα άλλο ερώτημα. Στο επόμενο σημείο τη σημερινή διάταξη θα πούμε ότι η θέση τη επιτροπή μα είναι ότι θα υπεραμεινθούμε τη θέσεω του προηγούμενου Κοινοβουλίου. Παρόλο που πολλοί από εμά δεν ήμασταν μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, είναι λίγο ασυνήθιστη αυτή η κατάσταση βέβαια, αλλά Κανένα δεν ξέρει κανένα, περισσότερο ε, πιο καλά τις, ε, τους κανόνες του Κοινοβουλίου από εσά. Εσείς τους συντάξατε. Εσείς τους γράψατε τους κανόνες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα, για να απαντήσω στη στήριξη των υπερπεριφερειακών περιοχών. Ε, Όντω, η συνθήκη έχει ειδικέ διατάξει για αυτέ τι περιφέρειες και τη στήριξη που πρέπει να του δώσουμε με συγκεκριμένα γεωγραφικά μειονεκτήματα. Για το μελλοντικό θα έχουμε προτείνει 350 εκατομμύρια ευρώ να δεσμευθούν για τη στήριξη αυτών των περιοχών. Επίσης έχουμε εισαγάγει μια διάταξη για ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα επιτρέπει σε αυτέ τι ε, υπεραπομακρυσμένες περιοχέ που εξαρτώνται από την αλία και θέλουν να διαφοροποιήσουν ε, και να περάσουν ας πούμε σε άλλε δυνατότητε όπω η ε, μπλε ανάπτυξη να μπορούν να το πράξουν. Τώρα για του καλού του κακού και του άσχημου, δεν θα σα πω εγώ ποιο είναι ο καλό, ποιο είναι κακό και ποιο άσχημος αλλά για το, σχετικά δηλαδή με το πώς δαπανούν τα κράτη-μέλη τα κονδύλια του ΕΤΘΑ αλλά όπως είπα και στην παρέμβασή μου στην αρχή, έχουμε κάποιες πολύ καλές ε, περιπτώσεις καλών πρακτικών και προσπαθούμε να τις ανταλλάξουμε ε, μεταξύ των κρατών μελών. Οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών συναντώνται σχετικά τακτικά για να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και να ενημερώνονται για νέες ιδέες, οπότε υπάρχει αρκετή ανταλλαγή που γίνεται σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του ταμείου, ποιε είναι οι προτεραιότητες και ποιε είναι οι καλέ πρακτικές. Τώρα, για το ερώτημα του κύριου Κόρμπετ ε, θα επιφυλαχθώ των ε, απαντήσεών μου για το επόμενο σημείο, μια που το ζήτησε και ο πρόεδρο. Για το ερώτημα τώρα για τα θαλάσσια απόβλητα, σίγουρα έχουμε δει ε, αύξηση στην τρέχουσα περίοδο, κυρίω τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, ε, στα προγράμματα αλλιεύω για απόβλητα. Α πούμε, ε, πληρώνουμε του αλλιεί να συλλέγουν απόβλητα ή να τα βάζουν σε ειδικέ αποθηκευτικέ μονάδε, είτε στο σκάφο είτε στο λιμένα, για να συλλέγονται τα απόβλητα αυτά. Είναι συνάδει αυτό και με την στρατηγική για τα πλαστικά που υιοθετήθηκε φέτο, όπου ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο για να βελτιώσουμε τα μέτρα που άπτονται της, ε, του αληφτικού κλάδου και της ε, συλλογή των ε, θαλασσιών αποβλήτων. Ελπίζω ότι έχω καλύψει τα πάντα, αν όχι ευχαρίστως να επανέλθω. Και βεβαίω θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το, για, το Ταμείο μετά το 2020 στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ για τι ευρύτατε απαντήσει σα. Οπότε πάμε τώρα στο σημείο 7. Να δούμε δηλαδή την κατάσταση για την νομοθετική ε, πρόταση για την ε, περίοδο 2021-2027. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2018, συζητήθηκε από την Επιτροπή μας την τελευταία θητεία και εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο λίγο πριν από τις ε, εκλογές, τον Απρίλιο. Ο Γκάμπριελ Μάτο ήταν ο εισηγητή μα τότε, ο οποίο δεν είναι εδώ. Αν γίνει το Brexit, βεβαίω θα εξαφανιστώ εγώ και θα εμφανιστεί αυτός, καταλαβαίνετε. Αλλά εν τω μεταξύ, ο κύριο Μιγιαμόν είναι ο εισηγητή μα. Παρακαλώ, σα ακούμε. Σας la situación, pero quiero... No, me parece que no va a depender ni de Γνωρίζω την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι δεν θα εξαρτηθεί η έκβαση ούτε από τον κύριο Μάτο, ούτε από εσά, ούτε από μένα. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται πολύ, σε επίπεδα πολύ μακριά από εμά. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον Καμπριέλ Μάτο. Πράγματι. Κατέβαλε προσπάθειες με διάφορου χειώδεις εισηγητέ, σημαντικέ προσπάθειε για να εγκρίνει το Κοινοβούλιο στι 4 Απριλίου, εάν δεν τα πατώμε, μια θέση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά ε, ισορροπημένη και θετική και θα αναφερθώ σε αυτήν αμέσω τώρα. Είναι η εντολή για να ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε εντολή είναι ένα σημείο εκκίνησης και ένας τριμερής διάλογος είναι μια ε, μακροχρόνια διαδικασία και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε τις αντίστοιχες μας θέσεις για να καταλήξουμε σε τελική συνένεση όλα τα θεσμικά όργανα και όλοι οι αρμόδιοι φορεί πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία αν πραγματικά έχουμε τη βούληση να καταλήξουμε σε συνένεση και σε συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο συνεχή με τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση σχετικά την περασμένη εβδομάδα, πολύ επικοδομητική κατά τη γνώμη μου και θα συνεχίσουμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Αφού μου το ζητήσατε, μου φαίνεται χρήσιμο να σας παρουσιάσω εν συντομία την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενστερνίζεται ένα μεγάλο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχιστεί η απλούστευση η διοικητική και να υπάρξει ευελιξία κατά την κατάρτιση και εκπόνηση των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η πρόταση της Επιτροπής και το περιεχόμενο της έκθεσης ζητά να ε, επιδιορθωθούν τα σφάλματα, τα λάθη. Είναι μια αρχιτεκτονική δομή πολύ περίπλοκη που μειώνει το βαθμό εκτέλεσης του προγράμματος μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον έτσι έχει συμβεί. Και ε, η αρχιτεκτονική δομή του ε, υπαρκτού προγράμματος, του υπαρκτού ταμείου, βασίζεται σε μια πολύ αυστηρή και άκαμπτη περιγραφή των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν και πρέπει να ε, εφαρμοστούν για να τύχουν ενίσχυση και χρηματοδότηση. Στη γραμμή λοιπόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ταμείο διαφαίνεται η φιλοδοξία. Εάν η χρηματοδότηση της επιχείρησης δεν περιγράφεται ρητός ως μη δυνάμενη, μη επιλέξιμη, τότε μπορεί κάλλιστα να συμπεριληφθεί. Δηλαδή υπάρχει πολύ πιο μεγάλη ασάφεια για το τι ενισχύουμε και τι χρηματοδοτούμε και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε μόνο κάτι το οποίο περιγράφεται ξεκάθαρα ως μη επιλέξιμο. Αυτό για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στο Ταμείο. Δεν είναι αυτός ο μακροσκελής κατάλογος απαρίθμησης ατελείωτων δράσεων ε, πολύ σαφώς περιγεγραμμένων οι οποίες ε, παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την ερμηνεία τους από τον εκάστοτε αναγνώστη. Και Στόχος είναι λοιπόν να ικανοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και να δοθεί ένα τέλος με τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει και δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας στόχος απλούστευσης αυτός που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό περιλαμβάνεται σαφέστατα στην εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει δηλαδή απόλυτη ταύτιση απόψεων επ' αυτού μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες αποχρώσεις έννοιες να έχουμε Φοροελία, προστασία των βιολογικών ε, πηγών, να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, της γαλάζιας ανάπτυξης, ε, με την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσες, στους ωκεανούς και ούτω καθεξής. Όλοι συμφωνούμε με το πρώτο σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε στην αηφορία των πόρων αλλά και στην κοινωνικο-οικονομική αηφορία και βιωσιμότητα. Και μιλούμε για τον στόλο, τον αλλιευτικό, τον τοπικό, τον τεχνικό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στα επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα σε εθνικό επίπεδο πρέπει να έχει ειδικό σχέδιο ε, δράσης, πρέπει να υπάρχει για τον ε, παράκτιο τοπικό αλλιευτικό στόλο. Και ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι η δεύτερη προτεραιότητα η υδατοκαλλιέργεια. Πριν από λίγες εβδομάδες μιλούσαμε για υδατοκαλλιέργεια στην ολομέλεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αλίας. Η υδατοκαλλιέργεια είναι σε τέλμα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ενώ αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμούς, με ρυθμούς στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ασκήσουμε ποιήση, να οθήσουμε, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά φάσης μεταξύ προσφοράς και ζήτηση στην Ευρώπη και θέλουμε να αυξηθεί η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους ε, του Ταμείου. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και ως εκ τούτου θέλουμε να λέγεται Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο Ταμείο Αλληλείας και Ιδατοκαλλιέργειας. Αυτό θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό συμβιβασμός. Οι ε, εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι άλλο θέμα. Ε, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κανόνες οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι στην, νομοθεσία, με συγχωρείτε εδώ και εκεί, ε, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλη η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διακυβέρνηση των ωκεανών, τη διαχείριση των ωκεανών. Δεν θα σας δώσω νούμερα ούτε ημερομηνίας, γιατί έχετε την εντολή γραπτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι διαθέσιμη για όλους. Λέγεται όμως το κείμενο ότι το 25% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κάθε κράτος μέλος θα προορίζεται στην αποκατάσταση της βιοπικιλότητας ε, στα θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και στην ε, θαλάσσια ερευνητική δραστηριότητα. Στην ερευνητική δραστηριότητα για αυτά τα επιστημονικά και θεματικά πεδία λοιπόν. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για την προστασία την αποκατάσταση της βιοπικιλότητας των οικοσυστημάτων, των θαλάσσιων και των παράκτιων. Υπάρχει και η στήριξη στην επιστημονική κοινότητα, στην συγκέντρωση δεδομένων για τον αντίκτυπο ε, στα πτηνά και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και η το επόμενο κεφάλαιο για την εντολή και για τη στήριξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Στην εντολή λοιπόν τη διαπραγματευτική που δίνει το Κοινοβούλιο απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα ουσίας και πρέπει τα κράτη-μέλη για το Κοινοβούλιο να δημοσιεύουν τις εκθέσεις τους για τις αιτήσει αποδόσεις. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ισορροπημένη, είναι μια πολύ καλή βάση για να διεξαχθεί αυτός ο τριμερής διάλογος επί τη βάση της συνένεσης. Ωστόσο θέλω να σταθώ σε δύο-τρία σημεία. Η διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θέλει ε, να πλήξει ε, τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τα ε, οικοσυστήματα. Ούτε θέλει τα λιευτικά σκάφη να αυξήσουν τη δυνατότητά τους να αλλιεύουν. Θέλουμε όμως παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν τις συνθήκες ασφαλείας και τις συνθήκες ε, ε, διαβίωσης των αλλιέων. Αναφέρεται άλλωστε στο άρθρο 13 αυτό. Μιλούμε για τα νέα σκάφη. Η εντολή του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει μόνο την ερασιτεχνική αλία και μετά υπάρχει αυτή η βασική αρχή που διαπνέει όλη την έκθεση ότι δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση της fishing capacity, της αλλιευτικής δυνατότητας. Άλλο η αύξηση του κινητήρα για λόγους ασφαλείας, για να μπορεί να πλεύσει το σκάφος στη θάλασσα και άλλο η αύξηση της αλλιευτικής δυνατότητας. Δεν σημαίνει ότι αυξάνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα πιο ευέλικτο καθιστός. Μιλούμε για τα σκάφη ερασιτεχνικής αλίας Ούτε σκοπός μας είναι να αντικαταστήσουμε κινητήρε με άλλους μεγαλύτερες υποδύναμεις. Θέλουμε να αποφύγουμε αρχαίους, πανάρχαιους κινητήρε που μολύνουν, που ρημαίνουν, να αποφύγουμε να παραμείνουν σε λειτουργία. ή ούτε θέλουμε να πλήξουμε τους αλληλείς με τις προσωρινές αναστολές αλλιευτικής δραστηριότητας. Όταν υπάρχουν αλλιευτικά ατυχήματα, να μπορούμε να επιβάλλουμε αυτή την προσωρινή αναστολή. Ή όταν υπάρχει ε, μία περίοδος ανα, ανάπαυλας για τον αλλιευτικό πληθυσμό, πρέπει να υπάρχει αυτή η αναστολή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κονδύλια τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά τα ταμεία είναι που επιτρέπουν την αναστολή και επιτρέπουν και τον παροπλισμό των πλοίων. Στόχος μας είναι να δώσουμε κονδύλια και στη γεωργία, δηλαδή να μην αυξηθεί η γεωργία τρίτων χωρών που μας πλημμυρίζουν με προϊόντα υποδέστερης και τελικά να μην έχουμε γεωργικά προϊόντα ευρωπαϊκά υψηλή ποιότητας. Αυτό που συμβαίνει στη Γεωργία λοιπόν δεν θέλουμε να συμβεί και στην Αλία να αυξηθεί η δραστηριότητα των τρίτων χωρών και να πλημμυρίσει τις αγορές μας με αλευτικά προϊόντα υποδέστερη ποιότητα. Υπάρχει λοιπόν αλευτικός κλάδο είναι σε καθυστέρηση, είναι σε υστέρηση και νομίζω ότι αυτά όλα που σας παρουσίασα συνθετικά απεικονίζουν την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαπραγμάτευση για τον τριμερή διάλογο. Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας με απλουστευμένες διαδικασίες, με αυξημένο προϋπολογισμό και αυτό είναι με στην εντολή ε, τη διαπραγματευτική. Αυτό θέλουμε εμείς για να καταφέρουμε και την ανανέωση των γενεών, να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η επόμενη γενιά θα πάρει τη σκητάλη Δηλαδή λένε πολλοί ότι θα μείνουμε χωρίς ψάρια στην Ευρώπη, αλλά εγώ λέω ότι θα μείνουμε και χωρίς ψαράδες. Και πρέπει κάτι να κάνουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για τα νέα μέλη, να σας πω λίγο τα διαδικαστικά. Η εκθεσία αυτή πέρασε από πρώτη ανάγνωση τον περασμένο Απρίλιο πριν τις εκλογές από το προηγούμενο κοινοβούλιο. Τώρα το συζητάμε στην Επιτροπή, θα, το ξανασυζητήσουμε, θα την ξανασυζητήσουμε στις 12 Νοεμβρίου όπου θα ψηφίσουμε κατά πόσο θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Τις τελευταίες 12 ημέρες πρέπει να έχετε λάβει εκατοντάδες email ε, και πάρα πολλά επαναλαμβανόμενα για αυτό το θέμα. Πολύ ενοχλητικό, ε, παρότι αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Ε, εκεί επισημανούνται κάποια θέματα. Ο κύριος Μιλαμόν είπε ότι οι προτεραιότητες μας είναι ίδιες με τις Κομισιόν. Είπε ότι μας απασχολούν οι κοινωνικο-οικονομικοί στόχοι, η βιωσιμότητα. Δεν θέλουμε περισσότερες δυνατότητες, ούτε υπεραλίευση. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν για ποιο λόγο ανησυχείτε για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολλές οι απαντήσεις για αυτό το ερώτημα. Δεν μας ανησυχούν μόνο οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Όταν κοιτάμε τις αντιδράσεις των ε, ε, συνομοθετών ε, ουσιαστικά λαμβάνουμε υπόψη και τις δύο θέσεις, όλες τις αντιδράσεις. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι γενικά, αλλά κάποια πράγματα μας δυσκολεύουν. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Χωρίς να πω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, το ζήτημα που μας απασχολεί περισσότερο και στις δύο θέσεις είναι το γεγονός ότι ανοίγουμε την πόρτα για κάτι που εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα επικίνδυνο η έννοια της ανανέωσης ούτε εξυγχρονισμού του στόλου. Θα το εξήγησα στην προηγούμενη μου παρουσίαση ότι το EMFF βοηθά τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική. Επίσης εξήγησα τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνουμε για να ασχοληθούμε με το ζήτημα της ανανέωσης των γενναιών, της ασφάλειας ε, ε, στον χώρο εργασίας, ε, της συνθήκες υγείας και ασφάλειας, ε, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κοινωνικο-οικονομικά μέτρα ε, για να ασχοληθούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως το Brexit, τη μία ανανέωση ε, συμπράξεων. Έχουμε πολλά τέτοια πράγματα τα οποία έχουμε συμπεριλάβει και στο προηγούμενο και στο σημερινό ταμείο για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα στα οποία αναφερθεί ο κ. Μιγιάνμον. Ωστόσο, μιλάμε για δημόσια χρήματα. Δημόσια χρήματα τα πρέπει να δημιουργήσουν συλλογικά, συλλογικά ωφέλη. Έχουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ενός ε, ε, παρκού επίπεδου διαβίωση για του αλληλεί, ε, τη συνθήκη ασφαλεία, να έχουμε επιστημιστική ασφάλεια κτλ. κτλ. Από την εμπειρία μας λοιπόν με την επανεισαγωγή των επιδοτήσεων για την ανανέωση ή την εξυγχρονισμό των σκαφών του στόλου αυτό ενέχει τον κίνδυνο κακών δαπανών δημόσιου χρήματος. Έχουμε κάνει πολλές αξιολογήσεις τις τελευταίες δεκαετίες που δείχνουν ότι οι επιβλαβείς επιδοτήσεις μπορούν και συμβάλλουν σε υπεραλίευση και σε υπερβολικές ελευτικές δυνατότητες. Κατά την άποψή μας το να ανοίξουμε το δρόμο για επιδοτήσεις όπως και να τις ονομάσουμε ανανέωση στόλου, εξυγχρονισμό σκαφών, αύξηση του ασφαλείας, ε, όλα αυτά ε, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Χαμηλή ε, προστιθέμενη αξία δημοσίων δαπανών, δημοσίων επενδύσεων. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για 22 μέτρα τράτα ε, πληρώνει κανείς 22 εκατομμύρια ευρώ. Ε, συγγνώμη, 3 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα δεκάμετρο πλοίο είναι 4.000 ευρώ. Έχουμε μικρό ταμείο, ορισμένα κράτη-μέλη παίρνουν μόλις 50-60 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δαπανίσουν σε 7 χρόνια για τη συλλογή δεδομένων, για έλεγχους, για υδατοκαλλιέργειες, για τοπική ανάπτυξη και για τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλία. Με αυτές τις τιμές λοιπόν ε, δαπανάς όλο σου το ταμείο με μια κίνηση. Η εκχώρηση κατά κράτο είναι 204 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αγοράσει 4 δεκατράτε με τόσα λεφτά. Σε ένα χρόνο τα προβλήματα τη δημοσιονομική εκτέλεση που αναφέραμε θα έχουν εξαφανιστεί. Οπότε επιστρέφω σε αυτά που είπα προηγουμένω, Έχουμε έναν τομέα πολύ επικερδή, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ του 2017. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία οικονομική αιτιολόγηση για επιδοτήσεις όταν υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις. Αν πάτε σε ναυπηγεία. Είναι γεμάτα με παραγγελίες για νέα σκάφη. Ήδη έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να αγοράσει ο τομέας και να εξυγχρονίσει. Δεν λέμε ότι δεν είναι δυνατόν. Φυσικά και μπορείς να το κάνεις. Αλλά μπορείς να το κάνεις με ιδιωτικά χρήματα και όχι δημόσια. Υπάρχει κίνδυνο δημιουργία τρευλώσεων στον κλάδο. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για όλου. Θα υπάρξουν συγκρούσει στον κλάδο μεταξύ όσων ε, παίρνουν χρήματα και όσων όχι. Και μετά συγκρούσεις και μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών, διότι τα μικρά κράτη δεν θα μπορούν να έχουν αρκετά χρήματα για να επιδοτήσουν έτσι τον αλληλευτικό του τομέα και έτσι θα δημιουργηθεί στρέβλωση στις θάλασσες μεταξύ των κρατών μελών που έχουν μεγαλύτερους στόλους και εκείνων που έχουν μικρότερους. Ξέρω ότι όλοι σας έχετε δεσμευτεί να διασφαλίσετε την κοινωνική βιωσιμότητα τομέα η ανανέωση των γενε... και την ανανέωση των γενεών στον τομέα Τη συνθήκες υγεία και ασφάλειας στον τομέα. Δεν το αμφισβητώ, αλλά το Ταμείο έχει αυτό το σκοπό ακριβώ, με την τρέχουσα μορφή του και όπως έχει στην πρόταση της Κομισιόν. Και αν οι συνομοθέτες επιμείνουν να ανοίξουν το δρόμο σε επιδοτήσεις για ανανέωση και εξυγχρονισμό στόλων, θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση ενώπιον τρίτων χωρών θα είναι αδύνατο να πούμε ότι έχουμε επιτύχει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, στο, το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 και ενδέχεται να δημιουργήσουμε μια κατάσταση σύγκρουσης δυσκολιών στον κλάδο για την οποία θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά που το κόμμα Brexit συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω βέβαια πόσο βοηθάει την καριέρα σας αυτό, κυρία μου. Ο κύριος Μιαμόν νομίζω ότι θέλει να απαντήσει. Θα έχετε την δυνατότητα βέβαια στο τέλος της συζήτησης. Οπότε να ακούσουμε τον εισηγήτη πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μετά τα όσα είπε ο κύριος Μινιαμών, θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δόθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. 497 υπερψήφισαν από τα 600 μέλη που πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Μεγάλη λοιπόν η πλειοψηφία. Βεβαίως το θέμα είναι περίπλοκο αλλά έχει γίνει και πολλή δουλειά για να μπορέσουν κάπως να συνδυαστούν, να συμφιλειωθούν όλες οι απόψεις. Πολλοί από όσου ε, ψήφισαν βέβαια δεν είναι εδώ τώρα, αλλά εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ε, βοήθησαν ε, και τους σοσιαλιστές και τη δική μου την ομάδα. Η συνάδελφος δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Το όραμα του ΕΤΘΑ είναι ότι θέλει να επιτύχει έναν αριθμό στόχων. Βεβαίω ε, η βιωσιμότητα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των θαλασσιών πόρων, των ωκεανών προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα, τα κονδύλια χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά, θα βοηθούν εκεί που χρειάζεται, τις ε, ε, ε κοινότητες, θα βοηθούν την μπλε οικονομία, την οργάνωση αυτής με καλύτερο τρόπο, προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα διάφορα κονδύλια που δίδονται από την κοινή αλληλευτική πολιτική, χωρίς βεβαίω να βλάπτουν, και αυτή είναι κόκκινη γραμμή, τους πόρους στους ωκεανούς, διαμορφώνοντας φυσικά και τις κοινωνικο-οικονομικές θέσεις μας για την αλληλεία. Οπότε η εντολή αυτή είναι πολύ καλή εντολή και είναι νομίζω κάτι που θα το δοκιμάσουμε στο διάλογο με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βιομηχανία, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά σίγουρα θα είναι μεγάλο λάθος εάν τα παρατήσουμε. Η εντολή αυτή, όπως είπα, ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά τελικώς επιτεύχθη με μεγάλη συνένεση. Αναφέρατε αυτά τα email που ξεκίνησαν να γεμίζουν τα inbox μας. Εγώ είμαι υπέρ, Πρόεδρε, του να συμμετέχουν οι πολίτες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ ήδη έχω πει και σε, στις ΜΚΙ ότι θέλω να ακούσω την απόψή τους. Δεν είναι ψηφιακή τρομοκρατία τώρα αυτή, δεν μας εμποδίζει σε τίποτα στο να έχουμε πρόσβαση στο email μας, επειδή είναι γεμάτο ας πούμε, και όπως ε, είπατε, ναι, και εμείς έχουμε εκατοντάδες email κάθε φορά που έχουν πάνω κάτω το ίδιο περιεχόμενο. Ε, προφανώς είναι μια απόπειρα lobbying αυτή, πίεσης. Αλλά αυτό γίνεται συχνά όταν προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπενθυμίσατε το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και ίσως το κείμενο όντως να εγκρίθηκε από την προηγούμενη Βουλή. Αυτό το δέχομαι. Όμως, το κείμενο το οποίο θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, δηλαδή το κείμενο που θα είναι αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου θα είναι ένα κείμενο που θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και θα γίνει αντικείμενο ψηφοφορίας του νέου Κοινοβούλου με τη νέα του σύνθεση. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να βγει από τον τριμερή διάλογο θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου και να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για το κείμενο που υιοθετήθηκε από το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Άλλοι αυτοί, άλλοι εμείς. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε στη, στη θέση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι, εν πάση περιπτώσει, μια ισχυρή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη χρηματοδότηση της γνώσης, στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Το 25% των κονδυλίων προβλέπεται από το κείμενο ότι θα στοχεύσουν προς αυτές τις επιδιώξεις. Να σταθώ όμως σε ένα σημείο, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Ταμείο δεν έχει άπειρες δυνατότητες, αλλά πεπερασμένες, 6 δις ευρώ. Πολλά είναι αλλά δεν είναι άπειρα και πρέπει να έχουμε πολύ σαφή και ακριβή στόχευση των ενισχύσεων των κρατικών, της κρατικής βοήθειας που δίδεται δηλαδή στον αλλιευτικό κλάδο, στον κλάδο της αλληλείας. Ο ωκεανός δεν έχει και τόσο μεγάλο βάθος δηλαδή τελικά. Υπάρχει το θέμα της προσαρμογής των σκαφών για την καλύτερη ασφάλεια, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων των αλλιέων και βεβαίως συμμεριζόμαστε την πράσινη συμφωνία, τον Green deal που η Επιτροπή Φοντεν Λάιεν θα μας παρουσιάσει ως ο νούπο. Άρα και η μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα από τα ζητούμενα. Συμφωνώ με τη συνάδελφο που ζητεί μεγαλύτερη ενίσχυση και ενσωμάτωση της περιφερειακής διάστασης που ζητεί περισσότερη περιφερειοποίηση. Ε, είναι μικρό το ταμείο και η Γερμανία δεν μπορεί να κάνει περιφερειοποίηση. Καλώς, αλλά η θέση στο άρθρο 9 του Κοινοβουλίου λέγεται ότι αν κάποια κράτη-μέλη θέλουν το κάνουν περιφερειακά. Αν όχι, επιθυμούν το εθνικό, επιλέγουν το, την εθνική άγουσα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει εμεί να παρέμβουμε στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα. Η περιφερειοποίηση είναι κλειδί για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδύλιων. Ε, κάποια στοιχεία πρέπει να μας ε, τραβήξουν την προσοχή και είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, με, όταν συναντηθήκαμε σκιώδεις εισηγητές με τον εισηγητή, ε, δηλαδή στο θέμα της δυναμικότητας, να μην αντιστρέψουμε την τάση. Μειωνόταν η δυναμικότητα με, τα τελευταία χρόνια και δεν πρέπει να ξαναυξήσουμε την αλευτική δυνατότητα. Και αυτό για διάφορους λόγους. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες σε ορισμένες αλληλευτικές περιοχές για να φτάσουμε τους στόχους της βέλτιστης επιτρεπόμενης απόδοσης έτσι ώστε να είναι πραγματικά βιώσιμη η αλληλεία. Άρα ας μην ξαναρχίσουμε με πρακτικές που είναι παν-αλλιευτικές και έχουν εξαιρετική δυνατότητα αλλίευσης και τα ε, μαζεύουν όλα. Έχουμε όμω και διεθνεί δεσμεύσει, οι οποίες μας λένε ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για μια βιώσιμη αλία στο σύνολο του πλανήτη, ξεκινώντας από, το, από τα του οίκου μας. Και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ε, υπενθυμίζοντας ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του ΠΟΕ. Δεν μπορούμε να, πηγαίνουμε λοιπόν στο ΠΟΕ και να ζητούμε από τις άλλες χώρες, από την Κίνα, από την Ινδία και το καθεξής, να καταργούν τις ενισχύσεις για την αυπήγηση νέων αλλιευτικών σκαφών, αν δεν πράττουμε και εμείς το ίδιο. Και το λέω γιατί είναι και οικονομικό το διακύβευμα. Αν και η Ινδία συνεχίζουν να ενισχύουν σκάφη που θα αλλιεύσουν σκάφη, ε, θα αλλιεύσουν αλλιεύματα, τα οποία θα καταλήξουν στα δικά μας πιάτα, γιατί εμείς είμαστε το 60 και 70% ε, των καταναλωτών των ε, αλλιευτικών προϊόντων τρίτων χωρών, ε, τότε αυτό που κάνουμε είναι να υπονομεύουμε τα θεμέλια του δικού μας σπιτιού. Ευχαριστώ, κυρία Κόντε, παρακαλώ. Αγαπητοί συναδελφοί, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στην προηγούμενη θητεία μας βρίσκει σύμφωνος γενικά. Θεωρώ σημαντικό κάποια σημεία να διαπρασπιστούμε περισσότερο από άλλα. Την αύξηση κατά 10% του προπολογισμού ε, τη θεωρούμε απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθήκων εργασίας, της ζωής, ε, την εκπαίδευση, τον κοινωνικό διάλογο και την αποσχόληση στον τομέα τη Η απλούστευση και σχετική πρόσβαση, ε, σχετικά με την πρόσβαση στο ταμείο πρέπει να είναι κατευθύνες γραμμές για να σχεδιαστεί ένα ταμείο το οποίο για χρόνια ήταν δύσκολο να εκμεταλλευτούν οι φορείς του τομέα. Η υπερβολική γραφειοκρατία συχνά είναι η βασική αιτία για την οποία υπάρχει, δεν, δεν δαπανώνται επαρκώς τα ταμεία. Υπάρχουν διάφορες δομές που μπορούν να διασφαλίσουν τις χρηματοδοτήσεις και επίσης χρειαζόμαστε τις ασφαλίσεις ε, σε περίπτωση περιστατικών ε, προβληματικών ή ατυχημάτων στη θάλασσα. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υποστηρίζει το μηχανισμός αυτός τους αλληλείς. Γι' αυτό το λόγο τα μέτρα που περιλαμβάνει πρέπει να ε, χαρακτηρίζονται από κοινωνικο-οικονομική υποστήριξη. Η προσωρινή μόνιμη πάυση, ο εξυγχρονισμός, η αγορά μικρής κλίμακα σκαφών και η αγορά νέων σκαφών με, χωρίς αύξηση όμως των ελευτικών δυνατοτήτων αλλά με μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ρήπανση είναι κάτι που υποστηρίζουμε με νέους κινητήρες ε, μετά από ζημιές που έχουν ε, προκληθεί από διάφορους λόγους ε, θα πρέπει να γίνει κάτι για τα ανεπιθύματα αλλιεύματα και άλλες και άλλα προβλήματα. Οι κυρώσει θα πρέπει να είναι πιο σαφείς, πιο λεπτομερεί. Οι αλληλείς πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Διαφορετικά θα του επιβάλλονται κυρώσει. Αν τους επιβληθούν κυρώσει, δεν πρέπει τα ποσά να είναι δυσανάλογα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδες ώστε στις 9 Νοεμβρίου να έχουμε μια κοινή ε, ε, εικόνα με την οποία θα συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία έτσι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την έκθεση αυτή. Η ανανέωση των γενεών, η αλληλεία, η υδατοκαλλιέργεια, συμφωνώ με τον κύριο Μιλανμόν. Υποστηρίξαμε την έκθεση αυτή φυσικά, αλλά έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Ορισμένα κράτη-μέλη λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από άλλα, κυρίως τα νέα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Κροατία, από την οποία έρχομαι και εγώ, είναι η χώρα μου. Θα ήθελα να επανέλθουμε στον κανόνα του νη Υπάρχει κάποιο σχέδιο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των ταμείων, γιατί είναι πολύ περιπλόκα. Η Κομισιόν βοηθά τα κράτη-μέλη απλουστεύοντας τα πράγματα. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου κάποια κράτη-μέλη έχουν τα ίδια περιπλέξει και δυσκολέψει περισσότερο τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Μια γρήγορη απάντηση από την Επιτροπή πολύ γρήγορα. Θα απαντήσω για δύο σημεία. Η ερώτηση της κυρίας Τόμασετς για τον Ίσιν 2. Όπως εξήγησα νωρίτερα, η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με τα κρατη για να προσδιορίσουν το μίσο που απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να επιταχυνθούν οι δαπάνες. Επίσης, είχαμε και την αναθεώρηση της απόδοσης φέτος. Τα κρατη εντόπισαν πού απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και έχουν ανακατανείμει ε, την χρηματοδότηση σε προτεραιότητες που έχουν καλύτερη απόδοση. Το άλλο με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε είναι κάποια άλλα σχόλια το ότι επενδύσεις για τα σκάφη και ο συγχρονισμός και η αγορά νέων σκαφών δεν αυξάνουν ε, λέτε ότι δεν αυξάνουν τη χωρητικότητα. Αυτό δεν συμβαίνει. Οποιαδήποτε επένδυση ανανέωσης εξυγχρονισμού σκάφους ή αγοράς σκάφους θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της αλληλευτικής δυνατότητας. Κατά κανέναν τρόπο δεν μπορεί κανείς να εξυγχρονίσει ένα σκάφος χωρίς να μπορεί αυτό να ψαρεύει περισσότερα. Γιατί? Διότι η κοινή αυξηση της αλληλευτικη δυνατοτητας κατα κανεναν πολιτική προβλέπει ότι η ικανότητα μετριέται σε ε, τονάζ σε όγκο δηλαδή και σε κιλοβάτ του κινητήρα. Και αυτό που ακούσαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας, οι συνάδελφοί μου από, την, από το τμήμα ελέγχου σας παρουσίασαν μια μελέτη για την επαλήθευση της υποδύναμης των κινητήρων. τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν επαληθεύουν σωστά την ισχύ των ε, κινητήρων, των μοτέρ. Δηλαδή δεν επαληθεύουν επαρκώς την ικανότητα του στόλου. Δηλαδή οποιασδήποτε επιδοτήσεις που ανανεώνουν, εξυγχρονίζουν, αυξάνουν την ασφάλεια, όπως και να το πείτε, θα αυξήσουν την ικανότητα, την ελευτική ικανότητα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να μπορεί να σχεδιαστεί από άνθρωπο που να έχει ως αποτέλεσμα μόνο εξυγχρονισμό ή ανανέωση χωρίς να αυξάνει τα ψάρια που πιάνει το σκάφος. Τα σκάφη γίνονται όλο και πιο δυνατά, πιο αποτελεσματικά, οι κινητήρες είναι όλο και πιο αποτελεσματικοί και με αυτό αυξάνονται και οι ελευτικές δυνατότητες. Μου λένε μερικοί ε, ε, με συγχωρείτε. Ήθελα απλά μια γρήγορη απάντηση για την κυρία Τόμασιτς. Ε, μια τελική απάντηση αυτό ήθελα. Ας το αφήσουμε εδώ και θα προχωρήσουμε. Κυρία Βούς. Ήθελα να πάρω το λόγο για να σας πω για το Ταμείο. Είναι τελείως αδύνατο αυτή τη στιγμή να δεσμευτούμε για την έναρξη τριμερούς διαλόγου. Έχουμε νέο κοινοβούλιο με νέους ερετούς. Ε, δεν μπορεί να κάνουμε τα ίδια σαν το παρελθόν. Υπάρχει αύξηση της αλληλευτικής προσπάθειας. Και για τους κινητήρες διαπιστώσαμε μαζική απάτη. 51% ήταν η απάτη στις διαπιστώσεις της προηγούμενης και οι επικουρικοί κινητήρες δεν ελήφθησαν υπόψη. Σε σχέση με τον Γάλλο συνάδελφο και τις διαπραγματεύσεις στο ΠΟΕ δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή γιατί θα αφαιρέσει αξιοπιστία από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Κόρμπερτ. Ευχαριστώ. Για τη θέση του προηγούμενου κοινοβουλίου που ίσως δεν είναι η θέση των νέων ερετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακόμα λιγότερο ακούγοντας τα πιστικά επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έπεισε ακόμα και τους οπαδούς του Brexit με την παρέμβασή της. Με ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος, όχι εσείς με ρωτήσατε. Ναι, αλλά μου, και δεν ξέρω. Ναι, αλλά μου πετάξατε πίσω το μπαλάκι. Επομένως, συνεχίζει ο βουλευτής, να σας ευχηστήσω την προσοχή στο κανόνα 61, ανανέωση παραπομπή στο Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου υπό το αίτημα της αρμόδιας επιτροπής θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπέμψει την πρότασή της ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Και μία από τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι ότι έχουν μεσολαβήσει εκλογές από τη στιγμή που υιοθέτησε τη θέση αυτή το Κοινοβούλιο. Επομένω, είναι ε, εφόσον θεωρεί ότι είναι αυτό επιθυμητό. Και βεβαίω είναι επιθυμητό όταν η άποψη του υφιστάμενου κοινοβουλίου φαίνεται διαφορετική από την άποψη του προηγούμενου. Ε, στην τρίτη παράγραφο ε, του άρθρου 7-8 έχουμε την επιλογή να αφήσουμε όλη τη διαδικασία και να έχουμε δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Στην παράγραφο 3 του 68 και όχι του 78, συγγνώμη, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε νέες τροπολογίες οι οποίες δεν επιδιώκουν μόνο απλό συμβιβασμό με το Συμβούλιο, αλλά νέες τροπολογίες εάν έχουν μεσολαβήσει κοινοβουλευτικές εκλογές εν τω μεταξύ. Είναι και ένας άλλος τρόπος να αναθεωρήσει το Κοινοβούλιο στην την υφιστάμενη του θέση για αυτό το αμφιλεγόμενο ζητήματα. Κύριε Κόμπεντ, αυτά που διαβάζετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που διαβάζω εγώ. Όμως ε, βοηθά την Επιτροπή να τα γνωρίζει όλα αυτά. Δεν τα διαβάζω το βράδυ, κύριε Πρόεδρε, στη δουλειά μου τα διαβάζω. Η κυρία Ντεμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. με τον κανονισμό για το περίοδο 2021 και 2027 έχουμε μεγάλη ευθύνη. Εγώ υποστήριζω το περιβάλλον, οπότε θεωρώ ότι έχουμε και μια ευθύνη για το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και για τους αλείς και για τους υδατοκαλλιεργητές. Θέλω να πω δύο λόγια για τη δυνατότητα που δίνει αυτό το κοινοβούλιο να παρασχεθούν χρηματοδοτήσεις για την αλλαγή ε, δραστηριοτήτων για μικρά αλλιευτικά σκάφη που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, το τονίζω. Εκεί οι νέα σκάφη μπορούν ενδεχομένως να αυξήσουν τα αλλιεύματα και δεν θα επηρεαστούν τόσο τα αποθέματα. Δεν, ε, η αλλία μικρής κλίμακας δεν επηρεάζεται τα αποθέματα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το είπατε και στην αρχή, ε, κυρία Σιγητά στη Μεσόγειο, αυτού του είδους η αλία επηρεάζει το οικοσύστημα πολύ μικρότερο από τα μεγάλα σκάφη ε, βιομηχανικής κλίμακας. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι ψαράδες ε, ε, ε έχουν, ε, δεν αντιστοιχούν παρά σε ένα πολύ μικρό κομμάτι των τοπικών εσόδων. Τα περισσότερα κράτη που ψαρεύουν στην Μεσόγειο χρησιμοποιούν σκάφη μέση ηλικία 30 ετών εκεί ούτε οι συνθήκες είναι αξιοπρεπεί, ε, οι συνθήκες εργασίας. Ας θυμηθούμε, ο Διεθνής Οργανισμό εργασία ε, και η Οδηγία 159 του 2017 δεν τηρούνται. Αλλά όχι μόνο αυτό, ε, τα σκάφη αυτά ρηπαίνουν. Χρειάζεται παρέμβαση σε τέτοιου είδου σκάφη ώστε να δοθεί μεγαλύτερη αξιοπρέπεια στους αλληλεί που καθημερινά εργάζονται σε δύσκολε και αβέβαιε συνθήκε, αλλά και για τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα που βλάπτουν τη βιομάζα των ωκεανών. Προφανώ η αγορά νέων σκαφών δεν πρέπει να επηρεάζει τη συνολική αλλιευτική ικανότητα ούτε να παραβιάζει τα όρια ισχύω των κινητήρων που προβλέπονται από του σημερινού κανόνε. Δικό μας καθήκον θα είναι να γίνει πιο ευέλικτο αλλά αποτελεσματικό το επόμενο σύστημα ελέγχων με κυρώσει ισότιμε και αναλογικέ, αναλογικέ με τι, με την, παραβίαση, με, την παραβίαση, με τον ψαρά που έχουμε μπροστά μα χωρίς να υπάρχει ε, κίνδυνος ε, να βλάψουμε ε, συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό το βλέπουμε στην Ιταλία αυτές τις μέρες. Υπήρξε μια έκθεση στην προηγούμε... του ελεκτικού συνεδρίου στην προηγούμενη θητεία όπου η Ιταλία δίνει δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι διότι παραβιάζει περισσότερο αλλά διότι ελέγχει καλύτερα τα πράγματα. Κάποιες παρατηρήσεις για τόσα είπε Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλά για την ανανέωση των σκαφών. Να αυξήσουμε λοιπόν τον προπολογισμό. Άλλη αντίρρηση, μιλάμε για δημόσιο χρήμα ε, που χρησιμοποιείται για έναν ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για την ΚΑΠ και για τους γεωργούς ε, και για όλους τους επιχειρηματίες. Ε, και αυτή η ιδιωτικοί τομέα είναι. Και αυτοί λαμβάνουν επιδοτήσεις και τις χρειάζονται για να προχωρήσουν, ειδικότερα σε περίοδους κρίσης. Τέλος, όλη αυτή η προσοχή που δίνεται ε, στα δημόσια χρήματα και με τόση ευχαρίστηση, αυτό το κάνει η Κομισιόν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι στην περίπτωση των μεγάλων πολυεθνικών, ε, και όσον αφορά τους αγωγούς φυσικού αερίου όλα αυτά τα οποία βλάπτουν το θαλάσσιο σύστημα και ρηπαίνουν. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε τον κατάλογο αγορητών τώρα. Επόμενος είναι ο... η κυρία Αγγιλέρα, παρακαλώ. Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι οι συνάδελφοι και σύντροφοι ήδη τα έχουν πει όλα και ο σκιώδης εισηγητής της πολιτικής μου ομάδας έδειξε τη θέση μας. Θα ήθελα να πω το εξής. Γνωρίζουμε τη θέση που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ερχόταν από καιρού καιρών ο κύριος Ματσάδο και μας την υπενθύμιζε. Μας υπενθύμιζε σε τι στραβό, πόσο στραβό ήταν ο δρόμος που είχαμε πάρει. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ερμηνεία. Εγώ δεν νομίζω και δεν πιστεύω ότι με αυτό που ενέκρινε εκπληρώνει το στόχο 14 της αηφόρου ανάπτυξης. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Είναι μια ερμηνεία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω και εγώ και η πολιτική μου ομάδα υπερασπιζόμαστε τις επιδιώξεις και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορεί κανείς να έρχεται εδώ και να λέει ότι αυτό που ε, ε, ενέκρινε το Κοινοβούλιο αντίκειται στο στόχο 14. Δεν συμφωνώ. Είναι δική τους ερμηνεία. Μία ερμηνεία μεταξύ πολλών. και υποτίθεται ότι δεν εκπληρούμε τα, τις προσταγές του ΠΟΕ. Και αν παραμείνει κάτι από το ΠΟΕ μετά τη διοίκηση Τραμπ, αυτό μένει να φανεί. Εγώ είμαι υπέρ της πολυμερούς ε, προσέγγισης. Και ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Το Συμβούλιο ήδη έχει ξεχωριστή θέση και το Κοινοβούλιο επίσης. Το είπε και ο Ρίτσαρντ. Όλα είναι δυνατά, όλα είναι εφικτά. Όλοι εδώ προδικάζουμε και λέμε ότι ίσως το νέο κοινοβούλιο δεν συμφωνεί ή μπορεί και να συμφωνεί. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν το έχει ερευνήσει κανείς και μεταξύ των βουλευτών ή δεν μου ζήτησε κανείς τη γνώμη μου τουλάχιστον, με ρώτησε αν συμφωνώ. Άρα πρέπει να προχωρούμε με βεβαιότητες. Με ανησυχεί αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε όλα είναι δυνατά και εφικτά. Αν είναι βούληση το, της πλειονότητας θα είχε φανεί. Κάνατε τη συζήτηση σε συντονιστές. Το κάνουμε ε, τη συζήτηση στην Επιτροπή. Λογικό είναι και καλώς να γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν μπορούμε να εκπέμπουμε εσφαλμένα μηνύματα στους πολίτες. Εάν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θα φανούν στις ψηφοφορίες και υπάρχει διαδικασία τριμερούς διαλόγου. Υπάρχει διαδικασία που τα εγγυάται όλα και που εγγυάται ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις μπορούν να απεικονιστούν και να αντικατοπτριστούν. Άρα, το μόνο που με απασχολεί είναι η εικόνα που δίνουμε προς το έξω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ολομέλεια. Και το λέω για να το ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει κάποιες επιφυλάξεις από ό,τι κατάλαβα για τη θέση του Κοινοβουλίου για την ανανέωση. Πώς θα το διαχειριστούμε προς το παρόν ακούσαμε από τα μέλη του κόμματος Brexit εδώ στην Επιτροπή ποια είναι η άποψή τους. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι θα πρέπει να καταστήσουμε πολύ το σαφές ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει δώσει πληροφορίες, απαντήσεις που ε, και κάποια κενά, γιατί η ανανέωση του στόλου είναι σίγουρα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα. Και επίσης έχουν ήδη ναυπηγηθεί και κάποια νέα σκάφη τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλά, πολύ αποτελεσματικά στην αλληλεία την οποία κάνουν και νομίζω ότι και αυτά θα συμβάλλουν στους στόχους της ελευτικής πολιτικής που είναι η επιλεξιμότητα. Είναι επίσης, ε, με, ε, χρησιμοποιούν υβριδικά καύσιμα και έτσι μπορούν να συμβάλλουν ε, στις ε, περιβαλλοντικές δράσεις και στόχους. Είναι περιβαλλοντικά φιλικά τα σκάφη αυτά και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γιατί να είμαστε αντίθετοι. Θεωρώ ότι αυτά ακριβώς, αυτοί ακριβώς οι είναι που χρειαζόμαστε. Και θα πρέπει να μπορούν να, χρηματοδοτηθούν από τον κορβανά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν είπε ότι ναι, αυτός είναι ένας ε, τομέας όπου πολλά ε, κονδύλια χρησιμοποιούνται και μπορούν να γίνουν και εξοικονομήσεις μέσω ανανέωσης, καινοτομίας, Α πούμε, τα... μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση από τα καύσιμα. Αυτά τα νέα σκάφη χρησιμοποιούν άλλου είδου καύσιμα. Εντάξει, κατανοώ αυτό που λέει και το κόμμα του Brexit, αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη όλα οδηγούν σε υπερδυνατότητα υπεραλίευση. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες οικονομι... ε, ε περιβαλλοντικές εξοικονομήσεις. Κάποιες από τις απαντήσεις της ε, Κομισιόν ε, δεν ήταν απολύτως ακριβείς. Και δεν μου αρέσει βεβαίω η αντίδραση του κόμματο Brexit, αλλά δεν μου αρέσουν και αυτά που λέει η Κομισιόν. Ο Ολλανδικό ε, στόλο είναι επικερδή. Ναι, αλλά όχι όλο. Γιατί, γιατί προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστο, το κόστο των καυσίμων και θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα, ε, επάρκεια στα καύσιμα. Εκεί αγγείται το όλο πρόβλημα στον Ολλανδικό στόλο. Η κυρία Οσάλιβαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις στη συζήτηση. Κάποια σημεία τα ανέφερε ο κύριος Μιγιαμόν. Αυτό που θέλω εγώ να πω και να σας επιστήσω την προσοχή είναι η έκθεση του ΟΗΕ για την παγκόσμια αξιολόγηση για τα οικοσυστήματα. Εκεί αναφέρεται ότι τα οικονομικά μέσα μπορεί να αποβούν ε, επιβλαβή στη φύση και περιλαμβάνονται εκεί επιδοτήσεις που κρύβουν το περιβαλλοντικό κόστος και υποστηρίζουν την μη βιώσιμη παραγωγή. Και έτσι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπεραλίευση και οι επιδοτήσεις για την αύξηση και τη διατήρηση των δυνατοτήτων πολλές φορές οδηγούν σε διάβρωση της φύσης. Επίσης υπάρχει και η έκθεση της Παγκοσμίας Τράπεζας που παρομοίω λέει ότι οι επιδοτήσεις μπορούν να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα και να διατηρήσουν την ανεπάρκεια. Επομένως υπάρχουν διάφορα σημεία στις εκθέσεις αυτές όπου οι επιδοτήσεις θεωρούνται επιβλαβείς προς τις αρχές της κοινή ελευθερικής πολιτικής, κυρίως ότι αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων και την ε, βιωσιμότητα. Και επίσης να θυμηθούμε και τον 14-6, το στόχο της βιώσιμη ανάπτυξης του ΙΕ, που λέει ότι οι επιδοτήσεις μπορεί να συμβάλλουν στην υπερβολική δυνατότητα, στην υπεραλίευση. Είναι στοιχεία που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Άκουσα τα όσα είπε ο κύριος Βαντάλεν. Και βεβαίω ότι σε ό,τι αφορά την ε, επάρκεια των ε, κινητήρων και την ισχύ τους πρέπει να καλωσορίζουμε την προσπάθεια που γίνεται να μην χρησιμοποιείται ας πούμε άνθρακας για, την, για ως καύσιμο, αλλά ε, εδώ υπάρχει και ένα μεγαλύτερο θέμα. Η διαφορά απόψεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσάνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχομαι από την Επιτροπή ΙΝΤΕ. Είμαι ε, εκπρόσωπο στο κοινοβουλευτικό, ε, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ. Και θέλω να πω ένα μήνυμα εδώ. Ανησυχούμε και εμείς ε, για την μεταρρύθμιση του ΕΤΘΑ που γίνεται θα ξέρετε σίγουρα εντός του πλαισίου του ΠΟΕ οι διαπραγματεύσεις για, για τον περιορισμό των επιδοτήσεων στον τομέα της αλληλείας είναι πάρα πολύ ε, δύσκολες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, προσπαθήσει να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μεγάλη κρίση στον ΠΟΕ και είναι πολιτικό, ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν επιτυχώς και έγκαιρα. Εάν τώρα το ΕΤΘΑ ε, μεταρρυθμιστεί σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου, ανησυχώ γιατί έτσι διακυβεύεται όλα, διακυβεύονται όλα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει την παραμικρή αξιοπιστία και πραγματικά δεν θα λαμβάνετε πια υπόψη από τους εταίρους της. Σας ενθαρρύνω λοιπόν αυτή την ε, οπτική να την έχετε υπόψη σας στις περαιτέρω συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Και ξέρω ότι παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφράσει και άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, θέλω να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Θέλετε το λόγο. Κύριε Βαντάλεν, δεν ακούσατε καθόλου τι είπα, γιατί θα έρθει μια μέρα που σίγουρα θα χρειαστείτε φίλους και θα καταλάβετε ότι πρέπει να, να τα έχετε καλά με το Ηνωμένο Βασίλειο όταν πάρουμε τον πλήρη έλεγχο των υδάτων μας. Οπότε όταν μιλάτε Μάλλον, αυτό που θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού φύγει και μετά, είναι βιώσιμη αλληλεία. Αυτό θέλετε κι εσεί. Άρα, εμεί θα μπορούμε να σα πούμε τι θα κάνουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Εμεί θα έχουμε σκάφη όχι πάνω από 25 μέτρα, όχι πάνω από 500 ύπου. Και αυτό πρέπει να αρχίσετε κι εσεί να το κάνετε, γιατί εσεί δεν θα έχετε τα μεγάλα σα τα σκάφη πια. Αν, έτσι, αν συνεχίσετε έτσι όπως μας επιτίθεστε, δεν θα έχετε ψάρια να πιάσετε, άρα δεν θα χρειάζεστε ε, σκάφη εμείς θα πάρουμε πίσω τα ψάρια μας. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βαντάλεν, θα, θα με χρειαστείτε ως φίλοι, προσέξτε το. Ευχαριστούμε. Ε, πάντα υπάρχει κάτι καλό στο τέλος κάθε κακού. Λοιπόν, συνάδελφοι, ήταν πραγματικά πολύ ωραία η συζήτηση. Ε, δεν, θα, δεν έχουμε κλείσει ακόμα, ως συζητητής θα πει τις τελευταίες του κουβέντες. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας δώσω και πάλι το λόγο. Ακούσαμε κάποιες ενσυχίες για τις ε, επιβλαβείς επιδοτήσεις, ακούσαμε τις απόψεις για τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν ε, σε ό,τι αφορά το, τη χωρητικότητα και την ισχύ των κινητήρων και οι διάφορες πτυχές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν όταν σχεδιάζουμε ας πούμε ένα νέο σκάφος και τι γίνεται με τους κινητήρες, ποιο σκάφος μπορεί να πιάσει περισσότερα ψάρια. Τούτων λεχθέντων, κανένα στην Επιτροπή δεν είπε ότι θέλει να αυξήσει τη δυνατότητα του στόλου. Δεν ακούστηκε κανέναν να πει ότι δεν θέλει να διατηρήσει τις αρχές της βιωσιμότητας. Όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τουαλέτες στα σκάφη, ότι τα συμφέροντα των μικρών αλλιέων θα προστατεύονται. Οπότε, γιατί εκφράζεται τόσες ανησυχίες για τη θέση του Κοινοβουλίου. Μήπω μπορείτε να πείτε κάτι τελευταίο πριν κλείσει ο κύριο Μιγιαμών. Um, Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι απλά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία θέση απέναντι στην οποία αντιδρούμε. Αντιδρούμε απέναντι στις δύο θέσεις και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διότι αυτά τα δύο θεσμικά όργανα μπαίνουν στη βασική τους φάση που είναι ο τριμερής διάλογος. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, δεν θέλουμε να αλλιεύουμε περισσότερο, θέλουμε να αλλιεύουμε καλύτερα. Λέτε πολλοί από εσά και συμφωνώ απολύτως. Και αυτό το ταμείο που φτιάχνουμε ακριβώς αυτό το σκοπό έχει. Περί αυτού πρόκειται και αυτό πρέπει να διαπνέει την οτροπία του. Όμως, Παραμένει το γεγονός ότι αν ανανεώσει κανεί τα σκάφη, αν τα εξυγχρονίσει, θα είναι πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και αυτό θα οδηγήσει σε υπεραλίευση. Πολλά σχόλια διατυπώθηκαν και λένε ότι έχουμε σύστημα ποσοστώσεων, μέγιστων, επιτρεπόμενων αλλιευμάτων και το καθεξής. Σας απαντώ λέγοντας ότι δεν καλύπτουν όλα τα αποθέματα. Σε πολλά είδη, σε πολλά ήχθη αποθέματα δεν έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης των αλλιευτικών ήχθη αποθεμάτων. Στην Μεσόγειο η ισχυρή πλειονότητα των αποθεμάτων υπεραλλιεύονται και αν ανανεώσουμε το σύνολο του στόλου αυξάνουμε την αλληλευτική πίεση και αυτό στα αποθέματα και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το λέμε ανοιχτά. Και τέλος, γνωρίζουμε καλά το θέμα ότι υπάρχει το ζήτημα με την ανανέωση των γενναιών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ζήτημα με τη γύραση του στόλου, με τις εργασιακές συνθήκες, με το ότι πρέπει να κατασταθεί ο κλάδος πιο ελκυστικός. Υπάρχουν πολλά κονδύλια στο Ταμείο για να τα καταφέρετε αυτά και η ναυπήγηση και ο εξυγχρονισμός των σκαφών δεν χρειάζονται για να προστατευτεί το εργασιακό δυναμικό ή να ανανεωθεί ή και να έρθει η νέα γενιά. Παρακαλώ να έχετε συνοχή στις απόψεις σας. Δεν μπορείτε να ζητάτε παροπλισμό αλλιευτικών σκαφών με δημόσιο χρήμα και άλλα χρήματα για προσωρινή αναστολή αλλιευτικής δραστηριότητας για να αντισταθμιστεί ο κλάδος από την άλλη και από την τρίτη πλευρά να λέτε θα αγοράσουμε και νέα σκάφη. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και λογοδοσία στον φορολογούμενο για το τι θέλουμε από το κλάδο μας και πώς τον στηρίζουμε. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τα, τις ερωτήσεις σας. Ήταν ένα πρωινό πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, για εμένα, στο οποίο ε, παρέστη με μεγάλη χαρά. Ο πρόεδρος, πολύ καλά τα πήγατε και ούτε νερό δεν σας φέραμε. Κύριε Μιγιάν Μον, έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου μιλητή. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν πολύ έντονη και παρατεταμένη η συζήτηση και δεν είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα που να ικανοποιούν τους πάντες. Να σταθώ σε δύο-τρία σημεία όμως και να προσπαθήσω να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι η θέση της ε, δεν, στρέφεται μόνο εναντίον του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου και βλέπει τα δύο θεσμικά όργανα να έχουν θέσεις τις οποίες δεν συμμερίζεται πλήρως. Θέλω να επαναλάβω την εξή ιδέα. Όταν γίνεται λόγος για ανανέωση του στόλου, για νέα σκάφη. Επιμένω, αυτά τα θέλουμε μόνο για την ερασιτεχνική ε, αλληλεία. Άρθρο 16. Δεν μιλούμε για νέα σκάφη γενικά. Μιλούμε για την, την αερασιτεχνική αλία μόνο. Και υπάρχει γενική αρχή η οποία στο άρθρο 4 λέει ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση δυναμικότητας, αλλιευτικής δυναμικότητας. Επιμένω όμως αγορά νέων σκαφών αφορά την αεραστεχνική αλία και μόνο. Και απαγορεύονται οι δεσμεύσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οι στόχοι με τις, ε, δεν ξέρω τι, με τις, ε, την αηφόρο ανάπτυξη κτλ. γίνεται λόγος. Το είπε η κυρία Γκιλέρα, ο στόχος 14 στο σημείο 6 δεν λέει ότι οι ενισχύσεις είναι όλες αρνητικές. Ενισχύσεις αρνητικές είναι αυτές που οδηγούν στην υπεραλήψη και στην υπερδυναμικότητα. Καταδικάζονται αδιακρίτω όλες οι ενισχύσει και επιδοτήσει. Άλλε είναι καλές όμως και άλλες είναι κακές. Και ε, με τις κακές ενισχύσει θα ασχοληθεί ο ΠΟΕ. Τώρα, Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Περσινή χρονιά, που επιτρέπεται σε δημόσια κονδύλια να αξιοποιηθούν για να νεωθεί ο αλλιευτικό στόλο στι εξόχω απόκεντρε περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να αναπηγηθούν δηλαδή νέα αλλιευτικά σκάφη και δεν είναι αλληλεία μέχρι 100 μέτρα βάθο, αλλά ε, πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή δεν ισχύει ότι ό,τι είναι δημόσιο χρήμα πρέπει να απαγορεύεται και είναι στρέβλωση της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επέτρεψε ειδικό καθεστώς για τη ρούπα για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες δηλαδή. Δεν θέλουμε να αλλιεύσουν περισσότερα τα σκάφη, θέλουμε να αλλιεύσουν καλύτερα και αυτό το λέει το άρθρο 3 για αυτό το οποίο είναι μη επιλέξιμο. Είναι τρεις ευρύ προϋποθέσεις. Εντός των ορίων του κράτους μέλους, εντό των ορίων τη αλληλευτική δυνατότητα του κράτου μέλου, χωρί να διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ της αλληλευτική δυναμικότητας και των δυνατοτήτων αλληλευτική δράση των υφιστάμενων, χωρίς να αυξηθεί και παραθέτω η δυναμικότητα, η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου αλληλευτικού σκάφους να αλλιεύει ηχθείες, θέματα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εισόδων και εξόδων, δηλαδή εάν ήταν αποτέλεσμα του εξυγχρονισμού να αυξηθεί η δυναμικότητα από τη μία, θα πρέπει αυτό να, να πέσει από την άλλη πλευρά. Αυτό το προσθέτει το Συμβούλιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον τριμερή διάλογο. Και ευχαριστώ τον κύριο Πισάρο. 494 ή 497 βουλευτές στήριξαν αυτή την εντολή με ελάχιστε αποχές. Είναι πολύ ευρεία η εντολή. Ξέρετε ότι το έχουμε ε, συζητήσει και στις συντονιστές. Η μεγάλη πλειοψηφία της, ε, ε, το ενέκρινε και η μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής το ενέκρινε. Εγκρίνει την εντολή. Να έχουμε πιο ευέλικτη θέση. Η θέση της Επιτροπής θα είναι πολύ σημαντική και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και θα φτάσουμε σε ε, συμβιβασμούς που θα σέβονται τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δεσμεύονται και τους στόχους μας για την αηφορία του περιβάλλοντος και για την κοινωνικο-οικονομική αηφορία. Τώρα, επιμένω, στον ΠΟΕ γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει δόγμα. Μία σειρά ενισχύσεων στο ΠΟΕ θεωρείται ότι δεν είναι αρνητικές οι ενισχύσει που έχουν να κάνουν π.χ. με την ασφάλεια του σκάφου και την ε, καλή διαβίωση των αλίεων. Να δούμε από χρώσε έννοιες. Αυτή τη στιγμή γίνεται διαπραγμάτευση για τελικό κείμενο στο επίπεδο του ΠΟΕ. Και ένα από τα σημεία όπου αποκλείεται η απαγόρευση των ενισχύσεων είναι οι ενισχύσει που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε τριμερείς διαλόγους με ανοιχτούς, επικοδομητικούς και η εντολή να εξελιχθεί και να προσωμιάσει στις θέσεις των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Και θα πρέπει τελικά το Κοινοβούλιο να ψηφίσει το αποτέλεσμα του τριλόγου και αν το κείμενο δεν μας ικανοποιεί δεν θα προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που έμαθα εδώ. Χρειαζόμαστε ένα κλάδο που να μπορεί να προσελκύει τους νέους. Οι βελτιώσεις στα σκάφη είναι χρήσιμες για τις συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας. Και τέλος. Ε, υπάρχουν όρια και κατόφλια. Η Λετωνία, η Ισπανία, η Πορτογαλία δεν μπορεί να πάρει όλα τα χρήματα και να τα ξοδέψει σε βελτιώσεις σκαφών και στον εξυγχρονισμό. Ό,τι έχει να κάνει με το εξυγχρονισμό δεν πρέπει να ξεπερνά το 60%. Δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια δεν ε, θα, δεν θα προωθηθούν για αντικατάσταση του αλευτικού εργαλείου. Ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο κοινοβούλιο όμως έδωσε εντολή και έχει ανανεωθεί κατά 60%. Οπότε υπάρχει μια δυνατότητα να δεχθούμε στην επόμενη συνεδρία στις 12 Νοεμβρίου τη θέση του κ. Κόρμπεν παρότι φανταζόμαι ότι θα δοθεί υποστήριξη για να συνεχιστεί η διαπραγματευτική θέση, όλοι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα το γεγονό ότι κανεί μα δεν θέλει να προωθήσει την υπεραλίευση ή να εισάγει επιδοτήσει που βλάπτουν το περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχουν ανεπιθύμητε Συνέπειε αν υποστηρίξουμε τη θέση του προηγούμενου κοινοβουλίου λίγο πριν τις εκλογέ. που ελήφθη λίγο πριν τι εκλογέ. Θα επανέλθουμε στην επόμενη συνεδρία και θα ψηφίσουμε ανάλογα. Προχωράμε τώρα και να ξαναευχαριστήσουμε την Κομισιόν. Πάμε στο σημείο 8. Υποψιάζομαι ότι μπορούμε, προλαβαίνουμε, έχουμε μόνο 10 λεπτά. Τέσσερι νέε ε, κατεξοδότηση πράξης που υιοθετούνται από το Κολέγιο των Επιτρόπων επιπλέον των τριών που εξετάζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μα αφορούν λεπτομέρειες υποχρέωσεων εκφόρτωση για ορισμένα βυθόβια είδη για την περίοδο 2020-2021 στη Βορειοθάλασσα, βορειοδυτικά υδάτα και νοτιοδυτικά υδάτα, λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίηση ε, διακοπής σε πραγματικό χρόνο ε, αλίας γαρίδας στο Σκάγκερακ. Τεχνικά σημειώματα, γι' αυτά θα σας στείλει η γραμματεία των συντομότερων δυνατών. Κομισιόν. Πού είναι η Κομισιόν. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά. Έχουμε χρόνο. Ή θα πρέπει να σας ζητήσουμε να επανέλθετε το απόγευμα. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις ε, έχετε. Δεν έχουμε καμία πληροφορία ακόμα όσον αφορά τα νέα κείμενα. Αν φιβάλλω να έχει κανείς ε, ε, να είναι σε θέση να κάνει ερωτήσεις κομισιών. Οπότε καλό θα ήταν να σας παρουσιάσουμε το περιεχόμενο των τεσσάρων της πράξεων των τριών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μία που αφορά την ε, Νορβηγία, αν συμφωνούν όλοι. Έχετε ένα λεπτό για το καθένα, για την κάθε της πράξη. Μπορώ να είμαι σύντομη, θα σας δώσω μια γενική εικόνα της προσεγγισής μας που μπορεί να σας ε, ε, χρησιμεύσει. Ξεκινάμε τις τρεις πρώτες της πράξης αφορούν ουσιαστικά τα σχέδια εκφόρτωσης για τη Βορειοθάλασσα, βορειοδυτικά υδάτα και νοτιοδυτικά υδάτα. βασικά για την υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Κάποιες πληροφορίες ε, το 2019 ήταν το πρώτο έτος πλήρους υλοποίησης των υποχρέωσεων εκφόρτωσης. Προφανώς αυτό είχε, ε, είχε συνέπεια δυσκολίες για το στόλο σε ορισμένες ελευτικές δραστηριότητες για να ασχοληθούμε με αυτές τις προκλήσεις. Η, η κοινή ελευτική πολιτική δίνει δύο οδούς, ε, για να το πω έτσι, για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η πρώτη είναι οι εξαιρέσεις ε, ε, σε περίπτωση υψηλή βιωσιμότητα, εφόσον υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο, υψηλού, υψηλά ποσοστά βιωσιμότητα. Το δεύτερο είναι οι εξαιρέσεις δε για περιπτώσεις όπου οι αυξήσει τη επιλεκτικότητα είναι δύσκολο να επιτευχθούν ή για τα αναλογικά κόστη ε, δυσανάλογα κόστη αρεπιθύμητων αλληλευμάτων. Αυτέ είναι οι δύο περιπτώσει. Σε αυτέ τι περιπτώσει, η Κομισιόν υιοθετεί κατεξοδότηση πράξη βάσει συστάσεων περιφερειακών ομάδων μετά από διαβούλευση με, με τι συμβουλευτικέ επιτροπέ. Θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να επιλέξει ίδια ό,τι θέλει. Ε, ακολουθούμε επιστημονικέ συμβουλέ του STCF. Είτε εγκρίνουμε είτε τα απορρίπτουμε. Δεν επιλέγουμε ότι μας αρέσει. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιηθήκαμε. Για αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια εκφόρτωση, οι κοινέ συστάσει εκπονήθηκαν κατά το πρώτο μισό του έτου. Πολύ δύσκολε συζητήσει στι περιφερειακέ ομάδε. Πολλά επιπλέον επιστημονικά στοιχεία, περισσότερα από ό,τι άλλα χρόνια. Λάβαμε τι τελικέ ε, κοινέ συστάσεις της 21 Μαΐου. Αμέσως εστάλησαν, υποβλήθηκαν μάλλον για αξιολόγηση στην STCF λάβαμε την εκθέση της STCF στα μέσα Ιουλίου και έκτοτε συζητάμε εντατικά με τις περιφερειακές ομάδες ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν τα δικά του σχόλια με τις επιστημονικές συμβουλές. Μια επιπλέον λεπτομέρεια στην παρουσιαφάση η Κομισιόν, αντίθετα από προηγούμενα χρόνια, ζήτησε από την STCF να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ειδικότερα για την εξοπιστία των σημερινών ερευνητικών προσπαθειών σε όλες τις περιφερειακές ομάδες την αναμενόμενη διάρκεια των ερευνών που τρέχουν και το κατά πόσο τα μέτρα επιλεξιμότητας ακόμα παίζουν ρόλο ε, για την επιλογή περτέρω μέτρων. Βάσει των συμβουλών της STCF, η Κομισιόν έλεγξε τις κοινές συστάσεις και έχουμε την ακόλουθη προσέγγιση. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της STCF ήταν θετική για μια συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε ναι. Αυτή είναι η εύκολη προσέγγιση. Το άλλο εύκολο σε περίπτωση που το STCF είναι αρνητικό για κάτι πάμε πίσω στις περιφερειακές ομάδες και τους ζητάμε να αφαιρέσουν τις δύσκολες περιπτώσεις που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικές συμβουλές. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα, αυτό συνέβη για τα νοτιοδυτικά ύδατα, όπου ζητήσαμε από την περιφερειακή ομάδα να άρει ε, για τρία ψάρια την εξαίρεση, το αίτημα εξαίρεση. Το ίδιο συνέβη και στα βορειοδυτικά ύδατα όπου δεν μας άρεσαν οι επιστημονικές συμβουλές για τα αποθέματα που υπόκεινται σε συμβουλή μηδέν ε, τάκα και σε κανόνες παράπλευρων αλλιευμάτων. Ε, τα αιτήματα δερμήνιμης που ήταν εκεί δεν μα άρεσαν γιατί πρόκειται για πολύ ευάλωτα αποθέματα και επιπλέον τον Ντεμίνιμι θα έθετε σε κίνδυνο περαιτέρω την κατάσταση των αποθεμάτων. Βγήκαν λοιπόν αυτά από την τελική έκθεση των ε, κοινών συστάσεων. Όπω είπα, η Κομισιόν δεν μπορεί να επιλέξει ότι τη αρέσει. Οι συζητήσει διέξαν πολύ καιρό με τι περιφερειακέ ομάδε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με τις ε, κατευθυντικές πράξεις ε, για να καταλάβετε ποια είναι η όλη εικόνα της διαδικασίας. Αλλά έχουμε πιστεί ότι στο τέλος της διαδικασίας αυτής ό,τι θα έχουμε μπροστά μας, την τελική έκδοση της κατευθυντικής πράξης, θα ευθυγραμμίσετε με τις επιστημονικές συμβουλές και με τις δικές μας ανησυχίες. Θα κλείσω εδώ να δώσω το λόγο στον συναδελφό που ασχολείται με τις συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Αυτή είναι η πρώτη κατεξοδότηση πράξη που προκύπτει από τον πρόσφατο κανονισμό ε, για τα τεχνικά μέτρα που πρόσφατα υιοθετήθηκε. Αφορά τη γαρίδα που ψαρεύεται στο Σκάγκερακ εκτενώς μεταξύ Σουηδίας, Δανίας και Νορβηγίας. Είχαμε πολλά παράπλευρα αλλιεύματα αγώνων και προτείνουμε ουσιαστικά ε, διακοπές ε, αλλιευμάτων σε πραγματικό χρόνο ώστε να αποτρέπεται ε, και απαγόρευση ορισμένων εργαλείων ώστε να προστατευθούν. Όπως είπαμε, τυσίως διαχειριζόμαστε εμείς με ΤΑΚ και η Νορβηγία. Το απόθεμα αφορά και τις δύο περιοχές, και ευρωπαϊκά έδατα και νορβηγικά. Ο σκοπός της κατεξουδότησης πράξης είναι η εναρμόνιση των τεχνικών κανονισμών που ισχύουν στα ευρωπαϊκά ύδατα, ώστε να συναδούν με τους κανονισμούς που ισχύουν στα νορβηγικά, τα σκάφη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο Σκάγκερα και υπόκεινται ε, στου ίδιου κανονισμού με αυτού που έχουμε στα νορβηγικά ύδατα. Να μην υπάρχει δηλαδή να έχουμε πλήρη κανονιστική ευθυγράμμιση και στι δύο πλευρέ του συνόρου, για να το πω έτσι. Ούτω ώστε τα σκάφη αυτά. Επιπλέον η κατεξοδότηση πράξη εισάγει δύο επιπλέον ιδιαίτερα επιλεκτικά εργαλεία για την προστασία των γονών που ονομάζονται για τα δύο ψάρια της περιοχής ε, ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει κίνητρο ώστε οι αλληλείς να χρησιμοποιούν επιλεκτικά, επιλεκτικά εργαλεία Αυτά ήταν τα βασικά ε, σημεία της κατεξουδότηση πράξης. Ευχαριστώ. Μπορεί να δημιουργήσατε τώρα κίνητρα για να τεθούν ερωτήσει, αν και δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια από τα μέλη. Να τα στείλετε παρακαλώ στην γραμματεία για να τα στείλει στην Κομισιόν και να μας στείλει γραπτό στις απαντήσεις της. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Είναι πάντα περίπλοκες αυτές οι εξαιρέσεις για τις ε, ε, υποχρεώσεις εκφόρτωσης και τις παρατάσεις αυτών. Θα τα συζητήσουμε όμως με περισσότερο χρόνο την επόμενη φορά. Ε, κυρία Βανέσκου, και ευχαριστώ και τον συναδελφό σα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στι 2.30. Έχουμε την έκθεση για την κατάσταση τη Μεσογείου που είναι πραγματικά καταστροφική. Έχουμε ένα σημείωμα για τα αποθέματα και τι περιοχέ ανάκτηση αποθέματο. Ελπίζω ότι θα ενδιαφέρει τον κύριο Μηγιαμό και την κυρία Αγγιλέρα αυτό, γιατί τα καλύτερα παραδείγματα περιοχών ανάκτηση είναι στην Ισπανία, μου είπανε. Δεν ξέρω. Οπότε φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει. Ελάτε παρακαλώ να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Και επίσης για το ε, ημερολόγιο σας έχουμε μία βραδινή εκδήλωση για την ε, αλληλή απλά, ε, που ελπίζω βεβαίω ότι θα παρευρεθείτε όλοι. Ευχαριστώ.